Dear colleagues, Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ομολόγους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε ξανά εδώ. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω τους ειδικούς προσκεκλημένους μας. Έχουμε δύο πρέσβεις εδώ σήμερα που εκπροσωπούν την ε, απερχόμενη Προεδρία, ο από πλευρά απερχόμενη ε, Προεδρία είναι ο κ. Ραϊμούντα Καρομπλή και η επερχόμενη Προεδρία, ο Θεόδωρο Σωτηρόπουλο, την εκπροσωπεί. Έχουμε επίση τον Επίτροπο, τον Ιωάννη Χάν, που όπω ξέρετε είναι ο υπεύθυνο Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική. Καλωσορίζω και όσου ε, έρχεστε εδώ για πρώτη φορά. Είναι η πέμπτη φορά που συνερχόμαστε στα πλαίσια της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εσείς ε, που έρχεστε στα Εθνικά Κοινοβούλια μας βλέπετε λοιπόν κανονικά για πέμπτη φορά, αλλά κάποιοι προφανώς έρχονται για πρώτη φορά και σας καλωσορίζουμε. Θα ξέρετε ίσως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια είσαστε εταίροι μας και όλοι μαζί εδώ και αρκετό καιρό έχουμε εμπλακεί ώστε να βρούμε την καλύτερη πλατφόρμα που θα εξασφαλίσει στη διαδικασία λήψη των αποφάσεων τη Ευρώπη μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα. Οι αιτήσει συναντήσει μα ήταν τμήμα αυτή τη διαδικασία, αυτή τη απόπειρα, ειδικά μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα, μέσω τη οποία ω κοινοβούλια έχουμε εξασφαλίσει μεγαλύτερε αρμοδιότητε, ακριβώ να γι' αυτό. Αυτή τη φορά θα εξετάσουμε τι προκλήσει για την εφαρμογή τη πολιτική συνοχή 2014-2020. Για μας ε, προκλήση σημαίνει και ευκαιρίες και προβλήματα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει ως βουλευτές να δούμε ποιες είναι οι ευθύνε μας πολύ προσεκτικά και να διαπιστώσουμε τι μπορούμε να κάνουμε ως εθνικά και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή ε, μέχρι το 2020 θα δώσει τα αποτελέσματα που αναμένουμε. Την περασμένη εβδομάδα στην Ολμέλεια του Στρασβούργου ολοκληρώσαμε μέσω της τελικής ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το κοινό μας έργο. Κοινό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπέβαλε την ε, πρόταση για το νέο ε, κανονιστικό πλαίσιο της ε, πολιτικής συνοχής και των δύο συνομοθετών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πολιτικής συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πλήρης ε, συνομοθέτης. Ε, οι, νομοθε... διαπραγματεύσεις πήραν πάνω από ένα χρόνο, ενώ έχουμε μπροστά μας για το μέλλον ε, το δευτερογενές δίκαιο το οποίο θα, το οποίο θα πρέπει να υιοθετηθεί με τη συνεργασία και των τριών θεσμικών οργάνων. Το αποτέλεσμα αυτού του διοργανικού διαλόγου και της προσπάθειας είναι μια, ένα πολύ καλό πλαίσιο πολιτικής συνοχής ε, που ανταποκρίνεται στις ε, ανάγκες του μέλλοντος. Ε, οι όλοι μας, ανεξαρτήτως της χώρας από την οποία προερχόμαστε, αναζητούμε ανάπτυξη, ανάπτυξη που θα βασίζεται σε καινοτομία, σε γνώση, σε αποτελεσματική χρήση των πόρων, ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας, μια ανάπτυξη που θα δίνει καλύτερη ποιότητα ζωής για μας και για τις επόμενες γενιές. Η, το επόμενο κύμα επενδύσεων που η πολιτική συνοχής άμεσα και έμεσα ε, μέσω της μόχλευσης ε, θα προσφέρει θα, ξεκινήσουν, ε, θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Οι στόχοι της νέας, της νέας πολιτικής καθώς επίσης και οι πόροι και οι επενδύσεις θα προχωρήσουν την Ευρώπη σε ένα δύσβατο μονοπάτι μέχρι το 2020. Δηλαδή η, η συνοχή, οι πόροι ε, και οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω των επενδύσεων. Στο πλαίσιο ισχυρών ανταγωνιστικών πιέσεων ε, και ελπίζουμε σε μια, μέσα σε μια Ευρώπη μετά την κρίση. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να γίνουν προγράμματα, επενδυτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των πόλεων, των περιοχών και των χωρών και σε εδαφική τοπική συνεργασία υψηλή προστέμενης αξίας. Μέσω της διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε τη δέσμευση να θέσει την πολιτική συνοχής ε, σε μια βάση ε, συνεργασίας. Θέλουμε να βελτιώσουμε την νομική ασφάλεια για όλα τα στοιχεία της πολιτικής και να αποφύγουμε ενδεχόμενες διαφορές στην ερμηνεία που θα δίδουν οι νομοθέτες, τα, οι νομοθέτες, τα κράτη-μέλη, ε, οι κομισιόν, ε, οι ελεγκτές και οι περιφέρειες. Προσπαθήσαμε να εξορθολογήσουμε την ερεσιμότητα, ε, εκ των προτέρων ερεσιμότητα και θα ήθελα να ε, ζητήσω και από εσά τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, να ε, ανδεσμευθείτε όταν εξαρτώνται από όταν εξαρτάται από εσά η εκ των προτέρων ρεσιμότητα να την χειριστείτε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα έτσι ώστε επενδύσεις να μην καθυστερούν εξαιτίας ε, καθυστερήσεων στα εθνικά κοινοβούλια. Αυτή η εκ των προτέρων αισιμότητα είναι μια ευκαιρία για να εντοπίσουμε νωρίς, όχι στην στιγμή του ελέγχου, ε, στην στιγμή του προγραμματισμού, ε, να εντοπίσουμε, λέω, εμπόδια στην εφαρμογή ή στην διενέργεια επενδύσεων. Οπότε εσείς στα Εθνικά Κοινοβούλια ζητούμε να εξασφαλίσετε ότι η εκ των προτέρων δεν θα ε, εμποδίζει αλλά θα βοηθάει το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής θα εξαρτηθεί από την ευρωπαϊκή διαδικασία διακυβέρνησης και ιδιαίτερα από το ε, ευρωπαϊκό ε, εξάμεινο και τις καταχώρασης συστάσεις. Τα εθνικά κοινοβούλια αποτελούν μέρος αυτής της διαδικασίας. Οπότε και πάλι σας ζητώ το εξής, να έχετε επαφές με τους συναδέλφους σας στις επιτροπές, που ασχολούνται με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Η καταχώρα συστάσεις όταν εφαρμοστεί αυτούν θα απαιτούν ε, συχνά ε, κρατικές επενδύσεις που θα χρηματοδοτούνται εν μέρη και από τα ταμεία συνοχής. Ε, αυτός ο, αυτός ο σύνδεσμος, αυτή η σχέση έχει συμπεριληφθεί στον κανονισμό των κοινών διατάξεων, σε αυτόν τον οριζόντιο κανονισμό και, και δείχνει πόσο σημαντική είναι η πολιτική συνοχή για τις επενδύσεις. Η σημερινή συνάντηση ε, θα έχει δύο τμήματα. Ε, σε κάθε τμήμα θα υπάρχει κάποιος που θα κάνει την εισαγωγή και μετά θα έχουμε ομιλητές και συζήτηση ε, μεταξύ τους. Οι ομιλητές προέρχονται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ελπίζουμε ότι θα δώσουμε 50 λεπτά για το διάλογο σε κάθε μία από αυτές τις δύο, δηλαδή σε κάθε μία αυτές τις δύο συνεδρίες. Παραδοσιακά έχουμε δύο ομιλητέ από τα Εθνικά Κοινοβούλια και έναν ομιλητή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά σειρά να εναλλάσσονται. Ορισμένοι από εσά έχετε δώσει τις ομιλίες σα. Ε, ε, ε, και έχουμε, μας έχετε δώσει τα ονόματά σας, όποιος άλλος θέλει να μιλήσει παρακαλώ να το αναφέρει. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την πρώτη συνεδρία Ε, καταρχήν ο πρέσβης Ραϊμούντας ε, Καρόμπλης που αντιπροσωπεύει την Προεδρία της Λιθουανίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα να, να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση. Ζητώ συγγνώμη που θα χρειαστεί να φύγω σχεδόν αμέσως μετά την ομιλία μου. γιατί πρέπει να προεδρεύσω στη συνάντηση του Κορεπέρ. Όχι για θέματα συνοχής, ούτε για θέματα ε, οικονομικά, αλλά για θέματα εσωτερικής πολιτικής. Η πολιτική συνοχή βρίσκεται στην καρδιά της προσπάθειας ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η βασική κριτήρια δύναμη στην αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επομένως, είναι υψηλότατη σημασία το γεγονό ότι την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πολιτική συμφωνία που επετέφθη στου τριμερεί διαλόγου για την τριμερή πολιτική στα πλαίσια του νομοθετικού πακέτου για αυτή την πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ μέχρι το τέλο του 2013. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ήταν μία από τις προσπάθειες και ένας από τους βασικούς στόχους της πρώτης προεδρίας της χώρας μου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά αυτό το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς ε, μεγάλη ευελιξία και από τους δύο συνομοθέτες. Θέλω να αναγνωρίσω τις προσπάθειες που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και οι συγητές που προσπάθησαν να καταλήξουν σε συμβιβασμούς. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερος την Πρόεδρο, την Τανούτα Χιούμπνερ, για την πολύ επικοδομητική προσέγγισή της. Τη στιγμή που οι θέσει των δύο θεσμικών οργάνων έμοιαζαν να είναι πολύ μακριά, καθώς και τον εισηγητή Φανίστερ Ρόι και τους υπόλοιπους σκιώδες εισηγητές ε, που βοήθησαν να συγκλίνουν οι θέσεις μας. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Χάν και την ομάδα του. Πιστεύω ότι χάρη στις προσπάθειες των τριών θεσμικών οργάνων, του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν, κάναμε καλή δουλειά. Μιλάμε σήμερα για ένα πακέτο κοινωνικής ε, πολιτική συγγνώμη συνοχή, ε, εξυγχρονισμένο, που να βασίζεται αποτελέσματα. Θέλω να επικεντρωθώ σε διάφορα νέα αποτελέσματα ε, που εισάγει το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και το πλαίσιο επιδόσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του μεταρρυθμισμένου πλαισίου, τη νέα προγραμματική περίοδο, είναι ότι συνδέεται άμεσα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη που να συμπεριλαμβάνει όλους. Μέσω του εισαγόμενου μηχανισμού της θεματικής συγκέντρωσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επικεντρωθούν ε, σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη στρατηγική του Ευρώπη 2020. Έρευνα και κοινοτομία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η χρηματοδότησή τους, ενεργειακή αποδοτικότητα, απασχόληση και κοινωνική ένταξη. Η τομεακή ε, εφαρμογή αυτό το, αυτής της θεματικής προσέγγισης θα διευκολυνθεί μέσω της νέας έννοιας του κοινού στρατηγικού πλαισίου που λαμβάνει υπόψη της, ε, την ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση και παρέμβαση από τα ταμεία που θα συμπληρωθεί με άλλα στοιχεία των ευρωπαϊκών πολιτικών και με διάφορα άλλα χρηματοδοτικά μέσα και μηχανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις από τα ταμεία δεν μπορούν να διαχωριστούν από τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Και αυτές οι ενωσιακές πολιτικές ε, στα πλαίσια του ορίζοντα 2020, ten μεταφορές δηλαδή για την ενέργεια, το Erasmus for Life κτλ. Και όλα αυτά πρέπει να, όλα να τα δούμε μέσα σε ένα ε, πλαίσιο. Θα υπάρξει καλύτερο συντονισμό μεταξύ όλων των πολιτικών και διαφορών επιπέδων ε, διαχείρισης. Θα υπάρξουν ε, περισσότερες πηγές χρηματοδότησης, θα δοθούν περισσότερες ευκαιρίες και θα είναι απλή η πρόσβαση για τους δικαιούχους. Θέλουμε ο ενωσιακός προϋπολογισμός να μην χρησιμοποιείται με άσχημο τρόπο, να μην υπάρχουν σπατάλες. Γι' αυτό οι συνομοθέτες ε, συμφώνησαν ότι το πλαίσιο επιδόσεων θα δημιουργηθεί για κάθε πλαίσιο, με σκοπό να παρακολουθεί την πρόοδό του προς την υλοποίηση των στόχων που έχουν ε, τεθεί για κάθε προτεραιότητα. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να θέσουν ε, πολύ φιλόδοξα ορόσημα και στόχους. Η εφαρμογή τους θα προσμετρηθεί στο τέλος της περίοδου προγραμματισμού. Το κανονιστικό πλαίσιο της νέας προγραμματικής περίοδου για την πολιτική συνοχή βασίζεται σε μια ισορροπημένη προσέγγιση και έχει μέτρα συντονισμού με σκοπό την ε, καλύτερη επίτευξη αποτελεσμάτων. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και πρέπει να δούμε ότι τηρούνται πριν χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια από τα ταμεία, καθώς και να αποθαρρύνουμε τις περιφέρειες από το να χρησιμοποιήσουν τα ταμεία με σπατάλες ή με ανεποτελεσματικό τρόπο. Μετά από ένα-δύο χρόνια διαπραγματεύσεων πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τις προσπάθειες και τα αποτελέσματά μας. Ε, ε, επενδύουμε σε εργασία και ανάπτυξη, όπως προβλέπει και η στρατηγική του 2020. Πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά πιστεύω ότι η διαπραγματευτική ομάδα που διαπραγματεύτηκε αυτό το αποτέλεσμα πιστεύει ότι οι προσπάθειες που θα γίνουν για επενδύσεις στον τομέα της απασχόλησης και της ε, ανάπτυξης θα είναι πολύ σημαντικές. Θέλω να συγχαρώ τα μέλη του Λιθουανικού Κοινοβουλίου η παρουσία του σήμερα δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα για τη Λιθουανία. Το 2010-2011 ήμασταν η χώρα με το υψηλότερο λόγο χρησιμοποίησης των κονδυλίων των Ταμείων Συνοχής. Μετά το 2009-2010 που είχαμε την κρίση, είχαμε μια ανάκαμψη των εξαγωγών μας. Και τώρα η εσωτερική κατανάλωση έχει αυξηθεί. Χάρη ακριβώς στα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής. έχουμε το υψηλότερο ε, ποσοστό χρησιμοποίησης, απορρόφησης των κονδυλίων των ταμείων συνοχής και πιστεύουμε ότι τα χρησιμοποιούμε πραγματικά αποτελεσματικά. Όλα τα κράτη-μέλη αυτό πρέπει να κάνουν. Οι περιφέρειες πρέπει να κάνουν ίσως περισσότερα για να καλύψουν το κενό που υπάρχει στην απορρόφηση των κονδυλίων από τα ταμεία γιατί μπορούν να αποτελέσουν προστιθέμενη αξία για την ε, δημιουργία θέσεων απασχόληση, για την ανάπτυξη και για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Μετά από μήνες συζητήσεων φαίνεται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στο να επιλύσει πολλά από τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Και λόγω της οικονομικής και χρηματοδοτικής κρίσης. Βέβαια αυτά τα, αυτά τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ και για την ψηφοφορία που είχατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Ο κύριος Σωτηρόπουλος, ε, εκ μέρους της Ελληνικής Προεδρίας, θα πάρει το λόγο τώρα. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή να είμαι μαζί σας σήμερα το απόγευμα. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω ιδιαίτερα τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η παρουσία τους δείχνει τις καλές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Και θα ήθελα να πω ότι είμαι ευτυχής για την παρουσία του Επιτρόπου Χάνα σήμερα μαζί μας, γιατί είναι κέρια η συμβολή του στην πρόθεση της πολιτικής συνοχής στα 28 κράτη-μέλη. Και τώρα, κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να περάσω στα ελληνικά. Ότι είναι θετικό ότι η, Ελλάδα λαμβάνει την προεδρία λίγο μετά από την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφίσεως κρίσιμων νομοθετικών πράξεων όπως οι κανονισμοί των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Οι βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας εγγράφονται απόλυτα στη λογική του νέου πλαισίου και επιδιώκουν να το αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ανάπτυξη και η απασχόληση, η εμβάθυνση της Ευρωζώνης, η μετανάστευση και η προώθηση της κινητικότητας καθώς και η θαλάσσια πολιτική, οι στόχοι δηλαδή της ελληνικής προεδρίας μπορούν να στηριχθούν αποτελεσματικά και να αξιοποιήσουν τις πολιτικές της νέας προγραμματικής περίοδου. Πριν προχωρήσω στην παρουσίαση των στόχων αυτών, θα ήθελα να υπενθυμίσω τις επίπονες διαπραγματεύσεις για την υιοθέτηση του νέου πλαισίου για πρώτη φορά συμφώνως με τις διατάξεις συνθήκης Λισαβόνας. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ο ρόλος των αρμοδίων επιτροπών του Κοινοβουλίου υπήρξε σημαντικός. Στον τομέα της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή Ρέτζι, οι επιμέρους εισηγητές, η πρόεδρος εσείς της Επιτροπής, αλλά και το σύνολο των μελών της λειτουργήσαν επικοδομητικά, εμπλουτίζοντας τις προτάσεις της Επιτροπής, συμπληρώνοντας ενδεχόμενες ατέλειες, ακόμα και διορθώνοντας ορισμένα σημεία προσαρμόζοντάς τα στις πραγματικότητες των κρατών μελών πάντα στη λογική των στόχων της Ευρώπης 2020. Με τον τρόπο αυτό το ήδη πολύτιμο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πλέον σε θέση να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Σήμερα και ενώ απομένει η ψήφιση ορισμένων ακόμα νομοθετικών πράξεων η Ένωση είναι σε θέση να περάσει στη νέα δημοσιονομική περίοδο εφαρμόζοντας τις πολιτικές του προγραμματισμού 14-2020. Είναι βεβαίως σε όλους μας γνωστό ότι το σύνολο του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως συγκρινόμενο με το συνολικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει περίπου το 1% σε όρους υποχρεώσεων και μόλις το 0,95% σε όρους πληρωμών χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα εκτός πλαισίου χρηματοδοτικά μέσα. Σε απόλυτο ωστόσο μέγεθος η Ένωση είναι σε θέση να επενδύσει την προσεχή επταετία σε τομείς και πολιτικές ε, προσανατολισμένες στο μέλλον ένα περίπου τρισεκατομμύριο ευρώ. Το μέγεθος αυτό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εφόσον γίνει η κατάλληλη αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στη σημερινή συγκυρία της κρίσης οι πολιτικές του νέου δημοσιονομικού πλαισίου είναι σε θέση να συμβάλλουν στην ανάκαμψη, στην τόνωση της απασχόλησης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η χρωματοδότηση του προπολογισμού της Ενώσεως είναι ακόμα πιο σημαντική τη στιγμή κατά την οποία η κρίση ε, αναγκάζει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν όλο και πιο σκληρές δημοσιονομικές πολιτικές. Είναι αλήθεια κυρία Πρόεδρε ότι η πολιτική της συνοχής αποτελεί την κατεξοχή πολιτική για τη στήριξη των επενδύσεων και την τόνωση της ανάπτυξης. Ο νέος τίτλος των διαρθρωτικών ταμείων, δηλαδή διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, αντανακλά, αντανακλά χαρακτηριστικά το στοιχείο αυτό. Η πολιτική της συνοχής στρέφεται πλέον ολοένα και περισσότερο από την στήριξη της υποδομής στη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στην περίπτωση πολλών κρατών μελών όπως και η χώρα μου η πολιτική συνοχής αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό επενδυτικό εργαλείο αλλά και μέσον για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Δεν θα πρέπει εξάλλου να αγνοήσουμε το γεγονό ότι η θεματική συγκέντρωση των πόρων των διαθετικών ταμείων με δεδομένο το ύψος των διαθεσίμων πόρων δίνει την δυνατότητα να διαμορφωθεί εκείνη η κρίσιμη μάζα η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικού αποτελέσματος. Στο πλαίσιο αυτό καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο περιβάλλον με την ικανοποίηση των εξάντε conditionalities, να τεθούν σαφείς αναπτυξιακοί στόχοι οι οποίοι μπορούν να ικανοποιούν τις απαιτήσει των κανονισμών έτσι ώστε μέσω της συγκέντρωσης των πόρων να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Οι προτεραιότητες έχουν, επιλογή, έχουν επιλεγεί με διάλογο σε όλα τα επίπεδα, έχοντας ως προϋπόθεση την επίτευξη μετρήσιμου και συγκεκριμένου αποτελέσματος. Από πλευράς μας θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για ικανοποίηση της απέτησης της προσθετικότητας, της additionality, απέτηση η οποία διευκολύνεται λόγω των ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για τα κράτα-μέλη σε πρόγραμμα. Στον τομέα της συνοχής θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο της υιοθέτηση της δευτερογενούς νομοθεσίας, εφαρμοσικές και κατεξιοδότηση πράξης, σε στενή συνεργασία όπως πάντοτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή. Επίσης, η Ελληνική Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ταχεία έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ταμείου Αλληλεγγύης εξυπακούεται ότι θα είμαστε σε στενή επαφή με όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου, την Επιτροπή και τους ε, λοιπούς οργανισμούς και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ολοκληρώνοντας, ε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ πολύ σύντομα σε ορισμένες εκδηλώσεις οι οποίες προγραμματίζονται από την Ελληνική Προεδρία στον τομέα σας. Πέραν της προναφερθήσης Υπουργικής Συνόδου, προγραμματίζεται συνάντηση ομάδας διαθετικών δράσεων στην Αθήνα στα τέλη Απριλίου. Επίσης προγραμματίζεται διάσκεψη για τη διαμόρφωση της μακροπεριφερειακής στρατηγικής Αδριατικής Ιωνίου, μία από τις προτεραιότητές μας, επίσης στην Αθήνα, μαζί με την Επιτροπή, στις 7 και 8 Φεβρουαρίου. Επίσης προγραμματίζονται και άλλες διασκέψεις και συναντήσεις όπως του Evaluation Network Group στην Αθήνα κτλ. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω ε, για την ε, ευκαιρία που μου δώσατε να απευθυνθώ σε ένα πάρα πολύ ε, σημαντικό κοινό και να ευχηθώ η επόμενη χρονιά να είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τις εκλογές μπροστά μας, να πάνε πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες να ψηφίσουν και να συνεχίσουμε σε έναν δρόμο στο οποίο θα κάνει την Ευρώπη πιο ισχυρή την Ευρώπη θα την κάνει με περισσότερες θέσεις εργασίας και με ακόμα πιο διαβριμένα τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη. Και χωρίς άλλο τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, δίνω το λόγο στον Επίτροπο Χάν. Ευχαριστώ Ντανούτα. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω θερμά. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική πρωτοβουλία αυτή, ότι σε τακτά διαστήματα έρχονται μέλη από τα Εθνικά Κοινοβουλία για ανταλλαγή πληροφοριών. Παρακολούθησα την εξέλιξη των γνωμοδοτήσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων επί νομοθετικών πρωτοβουλειών και βλέπω θετικότατες εξελίξεις από 168 το 67 σε 663 το 2012. Αυτό δείχνει ότι η αρχή της επικουρικότητας που εντάσσει στη λήψη των αποφάσεων τα εθνικά κοινοβούλια εντωμεταξύ έχει φάσει σε εντατικότατους ρυθμούς παρόλο που καμιά φορά γίνεται κριτική ότι όλες αυτές, όλες αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες υπάρχει όμως ένα θετικό ότι συμμετέχουν πάρα πολύ ένας μέγιστος αριθμός Καμιά φορά η δημοκρατία είναι χρονοβόρος διαδικασία, όμως δίνει την δυνατότητα να συμμετέχουν οι όλοι χωρίς ε, διαφοροποιήσεις και διαχωρισμούς. Ας αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται λοιπόν και για αυτές σας ευχαριστώ θερμά. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από διετής εντατικότατες διαπραγματεύσεις, για τις οποίες ευχαριστώ ιδιαίτερα την Ντανούτα Χιούμπνερ, του εισηγητές και τις διάφορες προεδρίες, που νομίζω συνολικά πέντε προεδρίες συμμετέσχουν. Ε, ειλικρινά όταν πρόκειται για την μελλοντική ε, χρήση των 325 εκατομμυρίων δίσε, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά και νομίζω ότι το αποτέλεσμα δικαιώνει τις προσπάθειες. Γιατί συνολικά μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε μια μεταρρύθμιση η οποία ίσως ε, ως προς την έκτασή της είναι η μεγαλύτερη μετά τη δημιουργία της περιφερειακής πολιτικής τη δεκαετία του 60. Αλλά αυτό ήταν πολύ σημαντικό, διότι έπρεπε να αντιδράσουμε στις εξελίξεις. Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε μέσα σε αυτό το διάστημα και η καθηγήτρια Χιούμπνερ είναι τώρα πρόεδρος της ε, Περιφερειακής Επιτροπής, αλλά υπήρξε και προκάτοχός μου επίτροπος και γνωρίζει όχι μόνο εξαιρετικά τα θέματα και μέσα από πολλά πρίσματα μπορεί να τα δει, αλλά και σε εκείνη και στην ομάδα της οφείλουμε το γεγονός ότι καταφέραμε να επιτελέσουμε πρόοδο και με την συνδρομή του Κοινοβουλίου, ώστε για πρώτη φορά να υπάρξει, αν θέλετε, μία σύνδεση των κονδυλίων προς συγκεκριμένους ε, στόχους ε, περιεχομένου. Δηλαδή υπήρχε σύνδεση προς τους στόχους της Λισαβόνας, υποχρεωτική για τα παλιά προαιρετικά για τα καινούργια και μπορούμε να πούμε ότι και για τις δύο ομάδες που έγιναν εντωμεταξύ μία, ε, ε, τα πράγματα πήγαν καλά. Τώρα προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα και είπαμε εντάξει, η περιφερειακή πολιτική είναι η καρδιά, αν θέλετε, των ε, πανευρωπαϊκών στόχων με αντίστοιχα οικονομικά κίνητρα και συνοδευτικά μέτρα και θα πρέπει να αξιοποιηθούν, να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη στόχων της Αναπτυξιακής Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Διότι ναι μεν ε, είναι ωραίο, αλλά είναι και πολιτικά πλοϊκό να πιστεύουμε ότι 28 κράτη-μέλη ταυτόχρονα θα επικεντρωθούν στους στόχους και θα προασπίσουν με την ίδια ε, επιμονή τους ίδιους στόχους και θα τους επιτύχουν και με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα με την ε, απαραίτητη προώθηση στις πολυάριθμες περιφέρειες της Ευρώπης να προωθήσουμε με διαφορετικούς ρυθμούς τους στόχους που είναι σημαντικό να επιτευχθούν για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Παράδειγμα, ε, αν ένας από τους στόχους μας είναι μέχρι το 2020 το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να το αυξήσουμε στο 20% της συνολικής παραγωγής ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση να την βελτιώσουμε ε, και την ενεργειακή επάρκεια, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις κλιματικές αλλαγές και την ε, προστασία του κλίματος, Πρέπει να λάβουμε κι άλλους εξίσου σημαντικούς παράγοντες υπόψη. Αν δούμε την δομή του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Ισοζυγίου θα λέγαμε ότι η Ευρώπη το 2012 μόνο στον τομέα των ε, ε, υπηρεσιών έχει πλεόνασμα 315 ή 317 δις μέσα από την εξάρτησή μας σε πρώτες ύλες, κυρίως πετρέλαιο και αέριο, αυτό το πλεόνασμα έγινε ένα πλήν 105 δις. Και βεβαίως ε, έχουμε εδώ την οικονομική διάσταση που μας δίνει τροφή για σκέψη, αλλά λέω ειλικρινά ότι αυτή είναι η αχίλιος πτέρνα της Ευρώπης, η εξάρτησή μας από πρώτες ύλες. Και αυτό το βιώνουμε οδυνηρά εν ώψη και των συζητήσεων για την Ουκρανία και τι επιπτώσεις θα έχει η εξάρτηση από τις προμήθειες πρώτων υλών. Πολιτικός μας στόχος πρέπει να είναι λοιπόν να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση με δεδομένο ότι ε, εμείς δεν έχουμε ευλογηθεί στην Ευρώπη να έχουμε πολλές πρώτες ύλε. Πρέπει λοιπόν να αντισταθμίσουμε αυτή την κατάσταση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο και ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές να επικεντρωθούμε εκεί και να, να, βελτιώσουμε την ενεργειακή μας ε, απόδοση. Ε, τα ενεργειακά κτίρια επηρεάζουν πολύ την ενεργειακή μας πολιτική και, αλλά και το εμπορικό μας ισοζύγιο σε τελευταία ανάλυση. Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους που θα βελτιώσουν και την παγκόσμια θέση μας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, γιατί Όσο λιγότερο εξαρτώμεθα από άλλους, τόσο ισχυρότερα, ισχυρότερη παρουσία έχουμε, όπου κι αν αναμειχθούμε στη διεθνή αρένα. Υπάρχουν αυτοί οι συσχετισμοί ορίζων 2020, δαπάνες για την έρευνα. Μια άλλη εξάρτηση της Ευρώπης ε, είναι οι σπάνιες γέες. Οι σπάνιες γέες χρειάζονται σε συγκεκριμένες τεχνολογίες ε, των ημιαγωγών για παράδειγμα, ούτω ώστε να παράγουμε διάφορα προϊόντα. Δεν μπορεί ως βιομηχανική περιοχή Ευρώπη να κάνει πίσω. Πρέπει λοιπόν να εισάγουμε σπάνιες γέες και σε αυτόν τον τομέα έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση. Πώς απαντάμε. Απαντάμε με ερευνητικά προγράμματα που σκοπό έχουν με τη βοήθεια βελτιωμένων τεχνολογιών να μειώσουν την χρήση την ποσότητα, της ποσότητας σε πρώτες ύλες ή με νέα υλικά και νέες εξελίξεις να παράγουν τεχνητές, πρώτες, ύλες που θα μειώσουν την εξάρτησή μας ή ε, θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα. Όλα αυτά γίνονται μόνο με κοινέ προσπάθειες και γι' αυτό η περιφερειακή πολιτική στο μέλλον συνεργάζεται στενά με τον ορίζοντα 2020. Ε, εδώ υπάρχει αυτό που λέμε brain circulation, γιατί στην Ευρώπη σε πολλούς τομείς έχουμε μεταναστευτικές κινήσεις όπου οι καλύτεροι μιας κοινωνίας μετακινούνται από μία περιφέρεια σε άλλες περιφέρειες. Η Λιθουανία μετά την προσχώρηση ε, η Λιθουανία έχασε το 10% του πληθυσμού της και μπορείτε να υποθέσετε ότι δεν ήταν χειρότεροι αυτοί. Από τη Ρουμανία έφυγαν εντωμεταξύ περίπου 2 εκατομμύρια και μετανάστευσαν σε άλλες χώρες για να απασχοληθούν εκεί. Πρέπει να προσπαθήσουμε με κατάλληλα μέσα λοιπόν από αυτήν την αφέμαξη, αυτό το brain drain, να κάνουμε κυκλοφορία εγκεφάλων, brain circulation. Ε, οι περιφέρειες μπορούν να μας υποστηρίξουν με θεματολογική επικέντρωση ε, για την επίτευξη στόχων. Με, αυτή, με αυτές τις εξάντε conditionalities που θα πρέπει να πληρούνται, ούτως ώστε τα χρήματα που διατίθενται να καταβληθούν. Διότι πάντα τίθεται το, η απέτηση να, χρησιμοποιείται με τρόπο να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια με τρόπο ποιοτικό όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται οι οικονομικές τους προοπτικές, η, οικονομική τους, το οικονομικό τους δυναμικό ή πού πρέπει να επενδύουν. Ή αν μια χώρα λαμβάνει κονδύλια για τον τομέα των υποδομών και τις μεταφορές, στο μέλλον τα επιμέρους προγράμματα δεν θα μας απασχολούν τόσο πολύ και αυτά, αλλά πρωτίστως θα μας απασχολεί η στρατηγική που αποτελεί τη βάση αυτών των επενδύσεων. Θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική συνολική των μεταφορών που περιλαμβάνει οδικές μεταφορές, σιδηροδρομικές, ε, ε, θαλάσσιες, ε, εναέριες. Ε, θα πρέπει να τα συνδυάζουμε όλα αυτά για να αποφασίζουμε εάν τα επενδυτικά μέτρα έχουν νόημα. Υπάρχουν λοιπόν στρατηγικές πάνω στη βάση των προγραμμάτων και όχι το αντίστροφο. Ε, σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ε, Περιφερειακή Επιτροπή ειδικότερα που φρόντισε να ε, θεσπιστούν ορισμένες κατώτατες τιμές, τιμές κατόφλια για την ενεργειακή επάρκεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν για διάφορους τομείς επενδύσεων. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος των εθνικών βουλευτών στον τομέα της εφαρμογής, της υλοποίησης. Τώρα διαπραγματευόμαστε τα προγράμματα με τα κράτη-μέλη και πολλές φορές εκφράζεται η επιθυμία για μεγαλύτερη ευελιξία. Και επιτρέψτε μου να πω ειλικρινά ότι καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι η ευελιξία ερμηνεύεται ως ελευθερία από τα πάντα. Η ελευθερία να κάνει κανείς τα πάντα. Έχουμε ε, υποβάλει έναν ε, μακροσκελέστατο κατάλογο. Τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να φτιάξουν με βάση αυτό τον κατάλογο ένα μενού πάρα πολύ δελεαστικό, αλλά παρακαλώ την κατανόησή σας. Ε, δεν υπάρχει δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε ιδιαίτερες επιθυμίες. Ε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο που πρέπει να ακολουθήσουμε και με τη βοήθεια των διαρθρωτικών ταμείων θα προχωρήσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται όμως στις διαπραγματεύσεις να προσέχουμε πολύ στην τήρηση των κανόνων του παιχνιδιού διότι το σημαντικό είναι οι πανευρωπαϊκοί στόχοι μας να επιτευχθούν μέσα από τις πολιτικές μας αυτές. Σε τελευταία ανάλυση προς το συμφέρον των Ευρωπαίων φορολογουμένων, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα λεφτά τους θα χρησιμοποιούνται με τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Περνάμε στους ε, δύο εισηγητές από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, καταρχήν ο Λάμπερτ Φανίστελροι Νίστελροι και μετά ο Γιάνν Όλμπριχτ. Ε, πέντε λεπτά στον καθένα δίνω μόνο. Ο κ. Βαν Νίστελροι. Χαίρομαι που βλέπω 15 συναδέλφους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης έτοιμους να ανταλλάξουν απόψεις με τους συναδέλφους των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Και το λέω γιατί η συζήτηση αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική στο Κοινοβούλιο. Πριν από πέντε χρόνια κάποιοι έλεγαν θα πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική συνοχή όπως την ξέρουμε και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις περιοχές Ευρωπαϊκής, περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα έπρεπε απλώς να δίνουμε λεφτά στους φτωχούς για να προσαρμοστούν. Και το αποτέλεσμα της συζήτησης τελικά ποιο ήταν. Ήταν μια μια νέα μεταρρυθμισμένη πολιτική συνοχής για όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για τις φτωχές περιφέρειες, με ένα, νέο συνδυασμό. Διότι είμαστε σε περίοδο εδώ κρίσης με μεγάλη ανεργία, απίστευτα νούμερα. Σε ορισμένες ε, χώρες ε, ε, ιδιαίτερα υψηλά. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να ξανασκεφτούμε τις αρχές πίσω από την πολιτική συνοχή. Η βασική αρχή τώρα θα πρέπει να είναι η συνοχή, η αλληλεγγύη, συγγνώμη, η αλληλεγγύη μεταξύ των πιο πλούσιων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, το, με τις αναπτυσσόμενες περιφέρειες. Και όπως είπε η Κομισιόν, δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι ορισμένες περιοχές της ε, Ευρώπης χάνουν τα πιο καλά μυαλά τους και τους νέους οι οποίοι μετακινούνται σε άλλες περιφέρειες Ευρώπης Ε, για παράδειγμα στην Πορτογαλία. Η πολιτική συνοχή δεν λειτουργούσε σωστά. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, ε, έχει πιο πολλούς αυτοκινητόδρομους κατά κεφαλή από τη Γερμανία. Και παρόλα αυτά 10.000 άτομα κάθε μήνα φεύγουν από την Πορτογαλία. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε την πολιτική συνοχή και το κάναμε. Δεύτερον, παρόλο ότι ε, οι εθνικοί ηγέτες είχαν ε, κάνει φοβερές, ε, πολύ ενδιαφέρουσες υποσχέσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής Λισαβόνας, να γίνουμε η πιο προηγμένη περιοχή του πλανήτη κλπ. κλπ. Δεν δούλεψε. Γιατί δεν... Κανένας δεν δέχτηκε να κάνει δική του τη στρατηγική Λισαβόνας. Οπότε έπρεπε να ξαναδούμε την ε, πολυεπίπεδη προσέγγιση. Αν η Ευρώπη θέλουμε να είναι πιο ευφυής, πιο οικολογική και να δώσει δουλειά στους πολίτες της, θα έπρεπε σε όλα τα επίπεδα ε, να υπάρξουν περισσότερες δεσμεύσεις, δηλαδή σε περιφερειακό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, σε κοινωτικό επίπεδο. Και αυτό έγινε μέσω της διαδικασίας ε, συνεργασίας, εταιρική σχέση την οποία εφαρμόσαμε. Και μετά, χρειαστήκαμε 80 τριμερείς διαλόγους. Ευρωπαϊκό ρεκόρ. Κακό ή καλό αυτό. Καλό. Γιατί τα κράτη-μέλη πριν από ένα χρόνο δεν ήταν έτοιμοι να δεχτούν κάτι διαφορετικό. Θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να συνεχίσουν όπως ήταν. Δηλαδή, να παίρνουν τα λεφτά και να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς όμως προωθούσαν μία, μεταμόρφ, αναμόρφωση. Και τώρα που ετοιμάσαμε τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, ε, θα χρησιμοποιηθούν για τα επόμενα 6-7 χρόνια για να εφαρμοστούν στρατηγικές των κρατών μελών. Και μετά έχουμε και την ευφύ εξειδίκευση. Τι είναι εφής εξειδίκευση. Είναι μια καινούρια έννοια με πολύ παρελθόν. Γιατί πολλά κράτη και πολλές περιφέρειες ακολουθούσαν τη δική του στρατηγική καινοτομία. Όμως μετά, αφού μάλλον η στρατηγική της Αβώνας ανέλαβε την ε, ε, πολιτική συνοχής, θέλουμε να συνδυάσουμε τις ε, περιοχές, τις περιφέρειες που έχουν συγκεκριμένη εξειδίκευση, συγκεκριμένη εμπειρία, για παράδειγμα νανοτεχνολογία, αυτοκινητοβιομηχανία κλπ. και να τις συνδέσουμε με πρωτοβουλίες αλλού στην Ευρώπη και να συνδυάσουμε έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση, βέλτιστες πρακτικές στις ε, επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τις μεγάλες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε αυτή είναι πλέον ε, εκ των προτέρων, δηλαδή πριν ξεκινήσει ο προγραμματισμός, κάθε κράτος μέλος πρέπει να προβάλλει, να ε, αποφασίσει ποια είναι τα δικά της project, δικές προτεραιότητες, τα κλάστερ της, ε, έτσι ώστε η ανάπτυξη να συνδυαστεί ε, σε όλες τις χώρες. Η στρατηγική Λισαβόνας απέτυχε και σήμερα αυτό που ζητάμε από τα μέλη του Ευρωπα... του... των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι να συζητήσουμε τις εθνικές κυβερνήσεις. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Γιατί δεν είναι κάτι που θα το προετοιμάσει ένας υπουργός ή ένα υπουργείο. Θα πρέπει να συμμετάσχουν οι πολίτες, τα πανεπιστήμια, η κοινωνία των πολιτών κλπ. Και μην ξεχνάτε ότι εδώ έχουμε και τον ορίζοντα του 2020 και την, την έρευνα, το πρόγραμμα LIFE και προφανώς και τα διαρθρωτικά ταμεία. Τελειώντας να πω το εξή. Έχουμε προσπαθήσει να καταλάβουμε ποια είναι η καινούρια πολιτική που χρειαζόταν και θα την εφαρμόσουμε τα επόμενα χρόνια. Ενδεχομένως ε, ξεκινάμε έτσι βέβαια, αλλά ίσως σε κανένα-δύο χρόνια θα πρέπει να δούμε τι έχουμε πετύχει και ελπίζω να έχουμε δει τότε τα αποτελέσματα μια κοινή πολιτική πιο εστιασμένη, πιο κοινή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταία εισαγωγή από τον Γιάνν Ολβιτ, που είναι η συγητής για το Περιφερειακό Ταμείο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είσαστε οι νομοθέτες και εμείς είμαστε νομοθέτες. Δουλεύουμε με διαφορετικά μέσα και μηχανισμούς. Εμείς σε αυτή την περίπτωση δουλεύουμε επί ενός κανονισμού. Όπως ξέρετε, ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ, σε εθνικό επίπεδο, χωρίς καμία άλλη διαδικασία εφαρμογής. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί τα Εθνικά Κοινοβουλία δεν ετοιμάζουν εφαρμοστικές πράξεις, καμία διαδικασία εφαρμογής για να εφαρμοστεί ο κανονισμός. Έχουμε τον κανονισμό γενικών διατάξεων και μετά έχουμε κάθε κανονισμό για κάθε ταμείο, όπως ξέρετε, για την πολιτική συνοχή. Ο, ο Μποστινάρο, ο Φανίστερόι, εγώ είμαι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, άλλος ε, για το Κοινωνικό Ταμείο και άλλος για το Ταμείο Εδαφικής Συνοχής. Εδαφική συνεργασία, συγγνώμη. Να πω κάποια στοιχεία από το κείμενο του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξη που πρέπει να εφαρμοστούν ε, σε επίπεδο κράτου σε διάφορα επίπεδα όμω στο κράτο. Καταρχά έχουμε τρία είδη περιφερειών. Όχι με τη διοικητική έννοια, αλλά σε επίπεδο ΝΑΤΣ 2. Λιγότερο ανεπτυγμένε σε μετάβαση και πιο ανεπτυγμένε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για κάποια κράτη-μέλη. Και έχουμε επίση τι περιφέρειες οι οποίες από λιγότερο ανεπτυγμένες έγιναν πιο ανεπτυγμένες, χωρίς να περάσουν τη διαδικασία με μετάβαση. Έχουμε περιφέρειες που είναι διαδικασίες, ε, περιφέρειες ας πούμε ε, σε ύφεση σχετικά, όπως τη Γερμανία, και τώρα είναι πιο ανεπτυγμένες. Κοιτάξτε προσεκτικά το κοινό, γιατί ανάλογα με τον ορισμό της περιφέρειας υπάρχουν ειδικέ προϋποθέσεις για κάθε μία από αυτές τις περιφέρειες. Μπαίνουμε στο είδος της ε, περιφέρειας. Το, το είδος της συγκέντρωσης εξαρτάται από το είδος της περιφέρειας. Άλλη συγκέντρωση για τις λιγότερο ανεπτυγμένες, άλλη για τις ε, περιφέρειες σε μετάβαση και για, άλλη συγκέντρωση για τις πιο ανεπτυγμένες. Για τις πρώην α, υπανάπτυκτες ας πούμε και τώρα ανεπτυγμένες είναι διαφορετική συγκέντρωση όπως ας πούμε για μια περιφέρεια στην Πολωνία ή κάποια από τα Λέντερ ας πούμε στη Γερμανία που δεν ήταν ανεπτυγμένα, αλλά είναι τώρα. Πρέπει να δούμε το επίπεδο συγκέντρωση. Από το 50% δηλαδή περνάμε στο 80% για δύο θεματικούς στόχους τουλάχιστον, δηλαδή καινοτομία, ε, πληροφορική, ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, μείωση των εκπομπών. Έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο ε, μείωση των εκπομπών για κάθε είδος περιφέρειας. 12% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες, αλλά αν μπαίνει και το Ταμείο συνοχή μπορούμε να πάμε πιο ψηλά. Για αυτές σε μετάβαση είναι 15% και για τις πιο αναπτυγμένες 20%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό το ποσοστό μπορεί να το ξαναδεί κανείς σε εθνικό επίπεδο, να αλλάξει δηλαδή σε εθνικό επίπεδο. Ε, είναι πολύ σημαντικό το είδο των επενδύσεων που θα είναι επιλέξιμε και στο κείμενο. Επί δύο χρόνια δουλεύαμε για να δούμε τα διαφορετικά είδη επενδύσεων που θα είναι επιλέξιμα. Να μην μπω σε λεπτομέρειε, γιατί πέντε λεφτά μου δώσατε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να διαβάσει κανείς πολύ προσεκτικά το κείμενο του κανονισμού για να δει πώς ερμηνεύεται το κείμενο. Τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να μπορούν να ερμηνεύουν το, σωστά το κείμενο. Οποιαδήποτε λάθη στην ερμηνεία των κριτηρίων επιλεξιμότητας θα, θα δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να δουλέψετε πολύ σκληρά για να καταλάβετε το κείμενο. Και το τελευταίο που θέλω να πω. Ε, μεγαλύτερος προσανατολισμός σε θέματα αστικά. Οι λεγόμενες βιώσιμες αστικές ε, δράσεις. Ε, τουλάχιστον 5% από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με ειδικέ προϋποθέσεις. Το ITI είναι η νέα μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί ε, στα ταμεία. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία της πολιτικής συνοχής. Είχαμε διάφορα προβλήματα. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η νοσιακή νομοθεσία στην ε, πολιτική συνοχή είναι τρομερά λεπτομερής. Δεν είναι μπλα μπλα όλα αυτά και φλιαρίες για το πόσο όμορφη είναι η Ευρώπη είναι τεχνικά πράγματα με πολλές λεπτομέρειες. Και χρειαζόμαστε μία μονοσήμαντη ερμηνεία. Όχι έτσι κι αλλιώ, Για να αποφύγουμε λάθη στην πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στου διάφορου στους διάφορους εκπροσώπους. Θα ήθελα όποιος ενδιαφέρεται να πάρει μέρος στη συζήτηση να μας πει τώρα, ούτως ώστε να ξέρουμε πόσο χρόνο έχουμε για τον κάθε ομιλητή. Γιατί αν ξέρουμε πόσο Ποιος είναι ο συνολικό αριθμό των ομιλητών, θα ξέρουμε πώς να διαρρέσουμε το χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν και οι εθνικοί βουλευτές και οι ευρωβουλευτές να μου πούν αν θέλουν να μιλήσουν. Ο κ. Βόλφκαν Χούμπερ, είναι από την Αυστρία και ο πρώτος ομιλητής. Τον Ευχαριστώ πολύ. Οι παρεμβάσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες ε, καλωσορίζω και τον Επιτροπό μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση στα Εθνικά Κοινοβούλια. Θέλω και εγώ να τονίσω αυτές τις ευκαιρίες που ανοίγονται στον τομέα της απασχόλησης και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Επίτροπος μίλησε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις, ιδιαίτερα εν ώψη της κρίσης, γιατί ε, ακούσαμε και μερικά παραδείγματα. Μιλήσατε για τους αυτοκινητοδρόμους στην Πορτογαλία. Και εγώ ξέρω ένα πολύ καλό παράδειγμα από την Ελλάδα, όπου περίπου 30.000 νέοι άνθρωποι ξαναγύρισαν στις ε, αγροτικές περιοχές, στην Ήπεθρο, για να στήσουν ε, μικρά, μικρές επιχειρήσεις δικές τους. Και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να αναφερθώ στις μικρές επιχειρήσεις. Και να αναφερθώ στη σπουδαιότητά τους γιατί ε, στα πλαίσια των επενδύσεων πολλές φορές θέλουμε να δράσουμε εξορθολογιστικά. Ο εξορθολογισμός μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερα στον γεωργικό τομέα. Ε, όταν η ανεργία είναι υψηλή και ρωτώ μάλιστα σε ποιο βαθμό στην παρακολούθηση της εφαρμογής και στα πλαίσια της συζήτηση ε, για τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης, σε ποιο βαθμό λοιπόν η Κομισιόν θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις όλων αυτών των συμφωνιών και λοιπά στην απασχόληση και θα προσδιορίσει ποσοτικά τη σημασία αυτών των προγραμμάτων, γιατί μου φαίνεται να είναι αυτό πολύ σημαντικό. Για το ρόλο των βουλευτών. Ε, ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Ως βουλευτής ε, που διαφοροποιείται και σε ένα περιφερειακό φόρουμ, θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου απλό να πιέσουμε τα αρμόδια καθήλυν Υπουργεία να ε, έρχονται στο Κοινοβούλιο και να ενημερώνουν για όλες αυτές τις εξελίξεις και προγράμματα, αλλά θα είχα μια πρόταση καλή. Θα ήταν μια ευκαιρία τουλάχιστον οι συμφωνίες εταιρική σχέσης να συζητούνται και να αποφασίζονται σε τελευταία ανάλυση και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήταν αυτό μια δυνατότητα, ούτως ώστε όλοι οι λεγόμενοι stakeholders, όλοι οι εμπλεκόμενοι από όλα τα επίπεδα να συμμετέχουν επαρκώς. Αν υπάρχουν προτάσεις από την Κομισιόν για το πώς θα δραστηριοποιηθούμε περισσότερο, ε, είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε και εμείς και να συμβάλλουμε. Ευχαριστώ. ο Άνδη Λούκας από, την, από τις κατοχώρες. Η Άννη Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση να έρθουμε σήμερα εδώ. Είναι σημαντική η ανταλλαγή απόψεων επί αυτών των θεμάτων με συναδέλφους άλλων χωρών. Και πριν αρχίσω την ομιλία μου θέλω να κάνω μια διαδικαστική παρατήρηση. Στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο ήθιστε να έχουν την ευκαιρία οι φιλοξενούμενοι να παίρνουν το λόγο πρώτοι. Ευχαριστώ που μας δώσατε την ίδια ευκαιρία και εδώ και θα ήθελα και αυτό το παράδειγμα να ακολουθηθεί και από άλλες επιτροπές και να ενθαρρύνετε τους συναδέλφους σας να ε, δίνουν το λόγο πρώτα στους ξένους φιλοξενουμένους τους και μετά στα μέλη του Κοινοβουλίου. Γενικά ε, το Ολλανδικό Κοινοβούλιο είναι ικανοποιημένο από τα αποτελέσματα στην πολιτική συνοχή και τις διαπραγματεύσεις και την ανάπτυξη και επιμερισμό της γνώσης. Αυτά χρειάζονται για να γίνει ανταγωνιστικότερη η Ευρώπη. Η κυβέρνησή μας ε, προσπαθεί να μειώσει τα κονδύλια διαρθωτικών ε, ταμείων ε, και τις επενδύσεις στην έρευνα ανάπτυξη. Το η Βουλή των Αντιπροσώπων χαίρεται διότι ο Ευρωπαϊκός Μακροπρόθεσμος προπολογισμό εστιάζει στην έρευνα και την ανάπτυξη και κάνει πιο στοχευμένη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Έτσι, η σχέση μεταξύ των δύο τομέων τη πολιτική αποκαθίστανται και οι περιφέρειες όλη την Ευρώπη μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη με βάση τη γνώση και ευχαριστώ τον συμπατριώτη μου τον κύριο Βανίστερ Ρόι που ε, κατάφερε ε, στις ε, μακρο, μακρές διαπραγματεύσεις να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να δημιουργούνται ευκαιρίες ε, να μην αντισταθμίζονται οι αδυναμίες. Ε, τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να μειωθούν ακόμη περισσότερο γι' αυτό. Ε, χαιρόμεθα για τις, και τις μακροοικονομικές αιρεσιμότητες και τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που περιλαμβάνονται εδώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που σεβαστήκατε και το χρονικό περιθώριό σας. Και τώρα από την Πορτογαλία ο κύριος Κάρλος Κωνστανέβες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είναι εξαίρετη αυτή η πρωτοβουλία που φέρνει κοντά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η Πορτογαλική Βουλή παρακολούθησε πολύ στενά την διαπραγμάτευση και θεωρούμε ικανοποιητικό το νέο πολιετές ε, πλαίσιο που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα πρέπει γρήγορα να περάσουμε στην πράξη, ε, να κάνουμε ε, λειτουργικό αυτό το πλαίσιο. Γιατί? Γιατί η ανεργία αυξάνεται, ιδιαίτερα η ανεργία των νέων. Το ίδιο και η φτώχεια. Και είναι αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν με την ιδεολογία που προασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την ε, απασχόληση, αλλά θα πρέπει γρήγορα να ξεπεράσουμε τη φάση της έγκρισης των προγραμμάτων ε, χρηματοδότησης χωρίς να περιμένουμε να λήξουν οι προθεσμίες. Τα επιχειρησιακά προγράμματα ε, δεν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2015 για να υλοποιηθούν. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε ήδη από το 2014. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να εξασφαλιστεί νωρίτερα. Και οι πολίτες θα πρέπει να αντιληφθούν αμέσως τα αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλειών. Εμείς από τη μεριά μας είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε να επιτευχθεί αυτό. Ευχαριστώ. Από Αντώνια Λάρκο από τη Γερουσία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για την ομάδα μας και για μένα τον ίδιο είναι τιμή που βρισκόμαστε εδώ. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μαζί με τον συνάδελφο Αντώνιο Ματσάδο. είναι σημαντικό που μας δίνετε ευκαιρία να εκφράσουμε την άποψή μας για τα, τις προκλήσεις ε, στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής ε, τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2020. Ε, αυτή εδώ η Επιτροπή είναι πολύ σημαντική και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας πιο στενά. Θα ήθελα να μιλήσω για τις ε, ε, περιφερειακές, εξόχως περιφερειακές περιοχές, απομακρυσμένες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ προέρχομαι από μια τέτοια και πιστεύω ότι η ειδική μεταχείριση αυτών των περιοχών θα πρέπει να αποτελέσει προϊόν μιας ισορροπίας που ε, οφείλεται στην, ε, στον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών των περιοχών θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τον όρο ε, άκρος ε, περιφερειακή συνοχή. Επίσης θα ήθελα να μιλήσω για την κοινωνική οικονομία στις ε, περιοχές αυτές. Ε, αν δεν μιλήσουμε για κοινωνική οικονομία δεν μπορούμε να μιλάμε για συνοχή. Πρέπει να προωθήσουμε την κοινωνική οικονομία ιδιαίτερα στιγμές που ζούμε. Άλλωστε αυτό ευθυγραμμίζεται και με τον ορίζοντα 2020, 2020. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο της φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Κίνδυνοι που είναι πάρα πολύ υψηλοί αφορούν 20 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή στις ε, άκρως απομακρυσμένες περιοχές, άκρως απομακρυσμένη συνοχή ε, και δέσμευση της Επιτροπής για την κοινωνική οικονομία και τον ορίζοντα 2020. Ευχαριστώ. Τώρα θα μιλήσει ένα ευρωβουλευτή, ο κύριο Αγκουράκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή όλες τις παρεμβάσεις και πρέπει να πω ότι ο κύριος Χάν ήταν για άλλη μια φορά αποκαλυπτικός. Ε, και από την τοποθέτησή του, αλλά νομίζω και από όλες αυτές τις συζητήσεις που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, υπάρχει ένα βασικό συμπέρασμα. Το βασικό συμπεράσμα είναι ότι δεν υπάρχει πλέον πολιτική συνοχής. Και καλό είναι να το πούμε αυτό το πράγμα. Τελείωσε η πολιτική συνοχής που ξέραμε δεν ενδιαφέρει πια κανέναν ούτε τυπικά εάν κάποιες περιοχές αναπτυχθούν πιο γρήγορα ώστε να φτάσουν σε ένα επίπεδο τις υπόλοιπες. Και επειδή βλέπω τον κύριο Βανίστερο να διαμαρτύρεται, θα τον ρωτήσω το εξή απλό πράγμα. Έχει υπόψη ο κύριο Βανίστερο τα επόμενα πέντε χρόνια ποια θα είναι οι διαφορές μεταξύ των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει γίνει κανένας υπολογισμός, έχει αποδείξει κανένας ότι τα προγράμματα για τα οποία μιλάμε πράγματι θα οδηγήσουν σε σύγκληση ε, των ε, περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει τέτοια μελέτη και ούτε μπορεί να υπάρξει γιατί, γιατί με τα προγράμματα αυτά θα υπάρχει απόκληση. Θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη απόκληση των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τους. Και θα υπάρχει αυτό για τον πολύ απλό λόγο Εξάλλου ακούσατε και τον κύριο Χάν. Ο κύριος Χάν μας είπε ότι το πρόβλημα της Ευρώπης είναι η ανέργεια και τα σπάνια μέταλλα, εν ε, Πώς θα γίνει όμως χώρες οι οποίες είναι πολύ χαμηλές στην παραγωγικότητα, στην παραγωγή, να αυξήσουν την παραγωγή τους. Και κύριε Βανίστερο, ε, αυτά που είπατε για την έρευνα και την βιομηχανία σε διάφορες περιοχές και να συνεργαστούν μεταξύ τους σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋπήρχε. Τα προγράμματα ΕΣΠΡΙ και τα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια υποτίθεται ότι αυτό θα κάνανε θα συνδέανε την έρευνα με την παραγωγή. Αλλά τι συνδέανε όμω. συνδέανε την έρευνα στι υπανάπτυχτε περιοχέ, όπου είναι φτηνή εργατική δύναμη, με την παραγωγή στι αναπτυγμένε και γι' αυτό κιόλα βλέπετε χώρε όπω η Ελλάδα, Πορτογαλία, η Ισπανία να, να αποκλίνονται και να φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ άλλε να αναπτύσσονται. Και με το πρόγραμμα αυτό που έχουμε, Ευρώπη 2020, αυτά τα φαινόμενα θα ενταθούν. Τελειώνοντα λέγοντα το εξή. Καλά, μπορούμε, μπορούμε βεβαίω να ειρωνευόμαστε τους δρόμους και ξέρουμε πολύ καλά ας πούμε ότι ε, στην Ελλάδα δυτικογερμανικές εταιρείες και γαλλικές εταιρείες έχουν ε, βγάλει μεγάλα κέρδη από δρόμους και μετρό. Όμως πριν τρει μέρες υπήρχε μια πλημμύρα στην, στη Ρόδο, πνίγηκαν τέσσερι άνθρωποι, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν υπήρχε δρόμος. Γιατί ο δρόμος έξω από την πόλη της, Ρόδου περνούσε μέσα από το ποτάμι. Και όταν ήρθε η βροχή δεν σταμάτησε η κυκλοφορία, πνίγηκαν οι άνθρωποι. Θέλω να πω με αυτό δηλαδή ότι αν στο παρελθόν έργα που έχει και ανάγκη ο κόσμος, αντιπλημμυρικά έργα, αντισυσμικά έργα, σχολεία, ε, ε, λαϊκή κατοικία δεν γινόταν γιατί δεν έχουν κέρδος, τώρα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα τα προβλήματα και τα προβλήματα ε, ε, ανεργίας, φτώχειας και αποκλεισμού που ζούμε αυτή την εποχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οξυνθούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Πάμε στο Δανέζικο Κοινοβούλιο. Η κυρία Ντέγκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου επιτρέπετε να παρέμβω στη σημερινή συνάντηση. Όταν συζητήσαμε για τα ταμεία και όταν τα συζητήσουμε στα διάφορα κράτη-μέλη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ένα μοντέλο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλες τις περιφέρειες, όλες τις περιοχές, και των πιο πλούσιων ακόμη κρατών μελών, γιατί και αυτά αντιμετωπίσουν προκλήσεις. Ε, έχουν τι ίδιε προκλήσεις όπως και οι περιφέρειε των φτωχών κρατών. Χρειαζόνται και εκείνε χρηματοδότηση με βάση το κατακεφαλήν ΑΕΠ Αυτό σημαίνει ότι τα φτωχά κράτη-μέλη στην προκειμένη περίπτωση έχουν ένα πλεονέκτημα, ενώ τα πιο πλούσια κράτη-μέλη αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Έχουν αστιφιλία, έχουν απερίμωση ας πούμε, των περιοχών της υπαίθρου, έχουν διάφορα προβλήματα και παρόλα αυτά με αυτό το μοντέλο που έχουμε προκρίνει δεν αποφελούνται καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν κάνω έκκληση όταν κάνετε τους υπολογισμούς σας για τη χρηματοδότηση να το κάνετε με βάση ένα μοντέλο που θα μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη τις γενικέ συνθήκες που υπάρχουν στις περιοχές της υπαίθρου. Εγώ θέλω ένα μοντέλο το οποίο θα υπολογίζει στις περιοχές της υπαίθρου τι επίπεδο ε, προσέλευση στο σχολείο έχουμε, ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής, ποιος είναι ο βαθμός αστικοποίησης, ποιος είναι ο βαθμός ε, απασχολησιμότητας. Ποια είναι αυτά τα ποσοστά, ούτω ώστε να βοηθήσουμε όλα τα κρατημέλη ε, και να τα αντιμετωπίσουμε πιο δίκαιο τρόπο. Όλα τα κρατημέλη που έχουν περιφερειακά προβλήματα ή ασδήποτε φύσης. Από την Τσεχική Δημοκρατία, ο Μίλος Βίστριτσινγκ από τη Γερουσία της Τσεχίας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Τσεχικού Κοινοβουλίου που μας προσκαλέσατε σε αυτή την συνάντηση. Άνω και κάτω βουλής εννοώ. Είμαι μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Γερουσίας. Και θα ήθελα να σας πω ότι όχι μόνο οι κυβερνήσεις, αλλά και οι περιφερειές μας εκπροσωπούνται εδώ. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι η εκ των προτέρων ερεσιμότητα είναι σημαντική για την αποτελεσματική περιφερειακή πολιτική. Το είπαν και άλλοι ομιλητέ, αυτό που είπε ο Επίτροπο Χάν, ότι θα πρέπει να έχουμε επαρκή χρόνο για να τα λάβουμε υπόψη όλα. Σωστό ίσω αυτό. Θα ήθελα να σας τονίσω ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε όταν προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε εταιρικέ συμφωνίες ε, οι οποίες δεν πήγαν καλά. Κάποιε από τι εκ των προτέρων προποθέσει, την αιρεσιμότητα δηλαδή, ε, συνδέεται με κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες που ενσωματώνται στην εθνική νομοθεσία. Αν η Κομισιόν δεν συμφωνήσει ότι αυτή ε, η ένταξη στην εθνική νομοθεσία έχει γίνει σωστά, τότε η Κομισιόν επιβάλλει κυρώσει σε αυτό το κράτο, ε, στο κράτο μέλο. Καταρχά, γράφει μια επιστολή προ αυτό το κράτο μέλο. Εν συνεχεία, θα πρέπει να απαντήσει το κράτο μέλο γιατί δεν περνάει στη σωστή εφαρμογή της ε, οδηγίας στην εσωτερική νομοθεσία και αν απαντήσει, ότι το κράτο, αν απαντήσει το κράτος μέλος ότι θέλει παράταση της προθεσμίας, τότε υπάρχει πρόβλημα για αυτό το κράτος μέλος. Το είπε και ο κ. Χάν. Και ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι η Κομισιόν δεν έχει προθεσμία ίδια για να απαντήσει επιστολές των κρατών μελών. Ας πούμε ότι έχουμε μια χώρα η οποία δεν εφαρμόζει σωστά μια οδηγία που συνδέεται με, τις με την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για θέματα, ας πούμε, ενεργειακής αποδοτικότητας. Ή παραδείγματο χάρη για καταναλωτικά κτίρια, ας πούμε, και ότι υπάρχει πρόβλημα την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων αυτών και το 2016. Εάν το κράτος μέλος δεν απαντήσει σωστά ε, στις ε, εγκλήσεις της Κομισιόν και αν δεν υπάρχει σωστή προθεσμία μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Ε, συζήτησα με τον κύριο Βλάσακ για να μου πει τι μπορεί να γίνει με τις προθεσμίες αυτές στην επαφή τους μέλους Κομισιόν. Γιατί αν έχει το κράτο μέλο προθεσμία για να απαντήσει, θα πρέπει η Κομισιόν να έχει αντίστοιχη προθεσμία, τέλο μια κάποια προθεσμία. Όχι να έχει ο ένα μόνο και όχι ο άλλο. Είναι πρόβλημα αυτό όταν διαπραγματευόμαστε τις ε, συμφωνίες εταιρική σχέσης. Ειδικά σε ό,τι αφορά την ε, συμμόρφωση με την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα. Ας πούμε ότι έχουμε ας πούμε, προθεσμία μέχρι το 2016. Αν η Κομισιόν όμως δεν έχει προθεσμία για να απαντήσει στις δικές μας απαντήσεις, τότε τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς γι' αυτό. Αν η Κομισιόν τρενάρει, ας πούμε, το πράγμα. Ευχαριστώ. Από την Ισπανία. Χωσέ Συζητούμε για την πολιτική συνοχής υπό το πρίσμα και μέσα σε μια συγκυρία βαριάς οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους πολίτες με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν χώρες που χάνουν, τα, μυαλά και άλλες που κερδίζουν. Υπάρχουν περιφέρειες και χώρες που θα αντιμετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες να συγκλίνουν προς, τον, προς τους ε, στόχους της ε, στρατηγικής 2020. Γιατί σημαίνει αυτό, γιατί αυτή η κρίση ανάγκασε τα κράτη-μέλη να ξαναρχίσουν να μιλάνε ε, για φτώχεια, για φυγή των νέων, για μαζική ανεργία κλπ. Ο Έλληνας εκπρόσωπος ε, μας μίλησε για αυτό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση με αλληλεγγύη και αλλοκατανόηση όποιοι είναι μακριά από την ε, συμμόρφωση, τη μακροοικονομική συμμόρφωση δεν θα πρέπει να αποκλειστούν. Ε, αν μπορέσουν να αποδείξουν ότι παρόλα αυτά κάνουν ό,τι μπορούν για την εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογία κλπ. όπως κάνουμε στην Ισπανία και στις ισπανικές περιφέρειες. Η Ευρώπη για την οποία πρέπει να στοιχηματίσουμε η Ευρώπη των πολιτών και των περιφερειών. Αν δεν είμαστε ικανοί να ερμηνεύσουμε την μακροοικονομική αιρεσιμότητα, οι διαφορές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα αυξηθούν το σημείο αφετηρίας είναι ότι ορισμένες οικονομίες, κυρίως της ε, Νότιας Ευρώπης, έχουν διαφορετική κοινωνική πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να μιλούμε για οικονομία μόνο με βάση ε, μακροοικονομικούς δείκτες. Θα πρέπει να μιλάμε για τους δείκτες ανάπτυξης, τη φτώχεια κλπ. Υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να αναρωτήσω τον Επίτροπο κύριο Χάν. Πιστεύετε κύριε Χάν ότι θα είναι δυνατόν να ή ερμηνευτεί η μακροοικονομική αιρεσιμότητα με τρόπο ευέλικτο, έτσι ώστε ε, μάλλον η ευελιξία για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης που ε, αντιμετωπίζουν τις δυσκολότερε συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ ο κ. Γιώζεφ Έκες από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Üdvözlöm a biztos Az Τα δυόμιση τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα και χρειάστηκε να δουλέψουμε πολύ για να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για τις προτάσεις της γιατί με βάση αυτές η Ουγγαρία θα έχει 35 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια στη διάθεσή της να ε, τα επενδύσει και ενώ η συγχρηματοδότηση πέρασε από το 75% στο 85%. Ε, δηλαδή 75% κοινοτικά κονδύλια, 15% ε, εθνική ε, συνεισφορά από το 75-25 που ήταν. Το 60% των κονδυλίων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επανεκκίνηση της οικονομίας και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ε, η ανεργία στην ε, Ουγγαρία έχει περάσει από το 4,5% στο 9,8%. Ε, η κεντρική Ουγγαρία αποτελεί μια περιφέρεια η οποία έχει δει την οικονομική κατάσταση να βελτιώνεται. και με τα καινούργια κονδύλια που θα μπορέσουμε να επενδύσουμε θα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την κατάστασή μας. Ε, θα αυξηθεί και ο προπολογισμό έρευνα και ανάπτυξης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, αντί για 16 προγράμματα θα έχουμε 9 μόνο στην Ουγγαρία. Το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν θέσει και το, ε, την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων ε, ως προτεραιότητα. Είναι πολύ θετικό, είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτό. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτά τα βήματα, βήματα τα οποία ε, δεν έχουν κάνει άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η τροφιμική ασφάλεια επίσης είναι προτεραιότητα για τις μελλοντικέ γενιές, για την επόμενη γενιά. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ε, μείωση των ε, περιφερειακών ανισοτήτων σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Να υπογραμμίσω το εξής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερη έμφαση στην δημιουργία επιστημονικών πάρκων καθώς επίσης και στην προάσπιση των ε, ευρεσιτεχνιών στην Ευρώπη. Ε, έχουμε μία μείωση του πληθωρισμού 0,9% τον Νοέμβρη ε, και ε, το έλλειμμα μας επίσης μάλλον θα είναι κάτω από το 3% στο τέλος του χρόνου. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε, τα αποτελέσματα έχουν έρθει, τα βλέπουμε ε, και αναμένουν τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ και συγχαίρω τον Επίτροπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο Γιώζεφ Ματούλα από τη Ρουμανία, Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος για να μην αναφέρω όσα ήδη ακούσαμε. Η νομοθετική δέσμη της επόμενης προγραμματικής περίοδου ε, επιτέλους εγκρίθηκε. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί και να εφαρμόζεται το συντομότερο δυνατόν για να αποδείξει την αποτελεσματικότητά της. Θα αναφέρω δύο θέματα που πιστεύω ότι είναι σημαντικά κυρίως για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. από τα συμπεράσματα των εκθέσεων προόδου 7 και 8 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την έκθεση για την εφαρμογή του Δημοσιονομικού Προγράμματος 2007-2014 μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση σταμάτησε τη διαδικασία σύγκλησης ή και την ανέστρεψε και οι ανισότητες μεταξύ περιφερειών έγιναν πιο μεγάλες. Έτσι ε, ε, τερματίστηκε μια μακρά περίοδος όπου οι ανισότητες μειώνονταν σημαντικά σε σχέση με το ΑΕΠ και την ε, ανεργία. Βέβαια με την κρίση επλήγησαν πρώτα οι πιο αδύναμες περιφέρειες. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα ε, εθνικά κοινοβούλια και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να εστιάσουν σε δύο τίνα. Ε, πρώτον, στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Εδώ θα ήθελα να με ενημερώσετε Πού έχουν φτάσει τα πράγματα με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, γιατί θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ την 1η Πρώτου του 2014. Οπότε χτυπάει ένα καμπανάκι σε σχέση με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Δεύτερον, ε, τα εναλλακτικά χρηματοδοτικά μέσα για μέσο και μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη είναι γνωστό ότι κυρίως στα νέα κράτη-μέλη η κρίση μπλοκάρισε όλα αυτά τα εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης. Αυτό το ομολογούμε, το λέμε και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι τράπεζες διασώθηκαν από την κρίση. Οι τράπεζες όμως και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι διατεθειμένα να βοηθήσουν να σωθεί και η οικονομική ανάπτυξη εκείνων των νέων, των νεότερων κρατών μελών μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα νέα κράτη-μέλη να βγουν από την κρίση. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό που πρέπει να μας απασχολήσει. Όπως ε, απασχολεί και τους εθνικούς βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ε, δημοσίευσε μια έκθεση που ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα. Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετέσχουν στην έγκριση αυτού του νομοθετικού πακέτου. Ιταλία τώρα. Ο κύριος Τομάσο Κόρο από την ε, Βουλή των Αντιπροσώπων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, διοργανωτές αυτής της διακοινοβουλευτικής συνάντησης, που είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να δούμε πού βρισκόμαστε στην πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η... Τα ταμεία για την πολιτική συνοχή είναι ένα σημαντικό ποσοστό του κοινοτικού προϋπολογισμού. Και γι' αυτό οι πολιτικές συνοχής έχουν ένα στρατηγικό χαρακτήρα στα πλαίσια των συνολικών πολιτικών που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως σε μια φάση όπου η έξοδος από την χρηματοοικονομική κρίση ε, αφορά πάρα πολλές χώρες. Σε πολλές χώρες υπάρχει δυστυχώς μια παρατεταμένη ύφεση, ακριβώς γι' αυτό υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ταμεία. Τα κονδύλια που υπάρχουν συνολικά για τις πολιτικές, με βάση τις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2014-2020, παρουσιάζουν μια μείωση 8% σε σχέση με την σημερινή περίοδο προγραμματισμού. Αυτό φυσικά δεν είναι θετικό. Η υπέρβαση των ανισοτήτων ανάπτυξης, η αύξηση το να υπάρχει ανάπτυξη γενικά, όλα αυτά είναι βασικά στοιχεία στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ιταλία, χώρα που μέχρι στιγμής μπορεί, παρουσιάζει τρομερές διαφορές ανάπτυξης ανάμεσα στο βορρά και στο νότο. Παρά επί πολλά χρόνια ήταν βασικός, ε, ε, μια από τις βασικές χώρες που συνεισέφεραν στον κοινοτικό προϋπολογισμό, δεν ε, υποφελήθηκε. Κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε πολιτικό και κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα κονδύλια των ταμείων και να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα. Προσπαθεί να βρει ποια είναι τα μέσα και οι μηχανισμοί για να αναπτύξει την παραγωγή της ε, και ποια είναι τα μέσα που πηγαίνουν για τις υποδομές. Και βεβαίως έχουν διαφορετική δυναμική τα μένα από τα δε. Η κυβέρνησή μας κάνει μια προσπάθεια υπευθυνοποίησης των τοπικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε και αυτοί να είναι σε θέση να ξοδεύουν καλύτερα τα κονδύλια που έχουν στη διάθεσή τους. Μέσω μια σειρά μηχανισμών που εισάγουν σε περίπτωση ανικανότητας να κάνουν κάτι τέτοιο, ε, την υποκατάστασή τους από τους εθνικούς φορείς. Δεν θέλουμε να υπάρξει διασπάθηση των πόρων. Θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα, ούτω ώστε να ενισχύσουμε τον παραγωγικό ιστό και την απασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μια σοβαρή ανησυχία που προκύπτει από, τις, από τον όρο της αιρεσιμότητας, κάτι που δεν υπήρχε στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Δηλαδή, για να υπάρξουν τα κονδύλια, θα πρέπει κάποια, κάποιοι όροι μακροοικονομικοί, στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης, να πληρούνται. Αυτό είναι προβληματικό. Και είναι προφανές ότι για μια χώρα η οποία βρίσκεται σε δυσκολία σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ε, μακροοικονομικών στόχων λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, εάν δεν υπάρχουν επιπλέον και τα κονδύλια από τα ταμεία συνοχή, θα σήμαινε ότι το μακροοικονομικό σενάριο του εν χωρας χώρα επιδεινώνεται φυσικά και μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο και μπαίνει σε μία ύφεση μετά από ύφεση μετά από ύφεση και είναι πολύ δύσκολο να κάμψει μια τέτοια χώρα. Εύχομαι λοιπόν να το ξαναδούμε αυτό το στοιχείο για να φτάσουμε σε πιο λογικές λύσεις για τις ε, χώρες μέλη που μπορεί να δείξουν και μία αποστροφή, μία απομάκρυνση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα λόγω αυτής της κατάστασης. Το σύμφωνο σταθερότητας ε, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι αυτά τα ταμεία θα πρέπει να αποτελέσουν ένα μοχλό ε, ολοκλήρωσης, ένταξης Αυτά που είπε δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε και ο Έλληνα συνάδελφο από, το... από την Ελληνική Βουλή. Το μιλητής εννοούσε προφανώ ο Έλληνα συνάδελφο απλώ. Ο επόμενος ομιλητής από την ε, Λετωνία. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που την ευκαιρία να πούμε την άποψή μας. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να εξασφαλίσει μια σταθερή ανάπτυξη των κρατών μελών. Και φυσικά τα ταμεία συνοχή είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ανάπτυξη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επικεντρώσουμε τους πόρους, να τους συγκεντρώσουμε και να τους δούμε σε αντιδιαστολή με τα αποτελέσματα. Προφανώς η εθνική χρηματοδότηση είναι απλή συγχρηματοδότηση. Δεν αρκεί από μόνη της, αλλά χρειαζόμαστε ένα σαφές σχέδιο που θα λέει ότι τα εθνικά, οι εθνικοί προϋπολογισμοί υποστηρίζουν και συμπληρώνουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τώρα, η χρηματοδότηση από τα Ταμεία Συνοχής υπάρχει για να εξασφαλίσει κάποια ισοτιμία, ας πούμε. Δηλαδή να επιτρέψει στους, πιο, στους λιγότερο ανεπτυγμένους να αναπτυχθούν και αυτοί προς τα πάνω. Φυσικά η μία λύση δεν είναι καλή για όλους, θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα εθνικά συμφέροντα κάθε κράτους μέλους και τις προτεραιότητες του κάθε κράτους μέλους. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου το κοινοβούλιο και η κοινωνία συμφωνεί ας πούμε, κάποια πράγματα, πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη. Εμείς στη Λετωνία έχουμε προβλήματα, έχουμε κοινωνικέ εντάσεις, αλλά δείξαμε ότι είμαστε σε θέση να ξεπεράσουμε την κρίση του 2008 και 2009, γιατί χρησιμοποίησαμε με συνετό τρόπο τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επόμενη τώρα περίοδο προγραμματισμού έχουμε αναπτύξει και εγκρίνει το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης από το Κοινοβούλιο είναι ένα έγγραφο προγραμματισμού που συνδέεται εκ του σύνεγγυς με τη στρατηγική του 2020. Σε αυτό το σχέδιο υπάρχει ένα στρατηγικό όραμα που βασίζεται σε μια λεπτομερή ανάλυση των βασικών αναγκών και των λύσεων που προτείνουμε. Επενδύσεις στις υποδομές. με σκοπό να έχουμε ε, μία μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν τα εθνικά συμφέροντα, το τονίζω αυτό, το υπογραμμίζω. Και ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνίε εταιρικέ σχέση, μάλλον στι διαπραγματεύσει για αυτέ τι συμφωνίε εταιρική σχέσει και να αρχίσουμε επιτέλου να χρησιμοποιούμε ε, αυτά τα κονδύλια από τα ταμεία έγκαιρα. Ο τελευταίο ομιλητή σε, σε αυτό το πρώτο πάνελ ο κύριος Πάντικ από την Κροατία, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι οι προηγούμενοι ομιλητές μίλησαν για τις μελλοντικές κατευθύνσεις που θα πάρει η πολιτική συνοχής ε, και έδωσαν έμφαση και στην ενεργειακή ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ, ερχόμενος από μια καινούρια χώρα, θα ήθελα να πω ότι οι προτεραιότητες μας εντάσσονται σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Η πολιτική συνοχής, κατά την μας, θα πρέπει να επηρεάζει την οικονομική πολιτική και τα οικονομικά αποτελέσματα. Συνεπώς θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια τα οποία αυξάνουν την απασχόληση και μας βοηθούν να αποφύγουμε την απώλεια των καλών μας μυαλών και εγκεφάλων. Τα διαρθρωτικά σχέδια θα πρέπει να οδηγούν σε οικονομική ανάπτυξη και σε αύξηση των θέσεων, επαρχία, ε, ε εργασίας. Τώρα, για την ανεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί ανάγκη για το μέλλον. Μία από τις δυνατότητες θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη και άλλων εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως το φυσικό αέριο. Η Κροατία ε, ετοιμάζει στο, στην Ίσο Κέρκ ένα, ε, ένα τερματικό σταθμό ε, φυσικού αερίου και θα μπορούσε να, αυτό να αποτελέσει μια εναλλακτική οδό και για την Κροατία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο από τη Ρουμανία, ο Πέτρο Λουχανέκ, εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Δράτω με τις ευκαιρίες, μια και έχουμε τον Επίτροπο και έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε για την πολιτική συνοχή με τους αξιότιμους εθνικούς βουλευτές, να πω ότι έχουμε κάποιες κοινέ γραμμές πλεύσης εδώ Άκουσα πολλά για τις πιθανές επιπτώσεις και από τους γερουσιαστές και από τους βουλευτές τους εθνικούς αλλά θεωρώ ότι μιλήσαμε λίγο για τα αίτια π.χ. γιατί το ποσοστό απορρόφησης στις περιφερειακές χώρες είναι τόσο χαμηλό. Στην πατρίδα μου, τη Ρουμανία, για παράδειγμα, ε, η κατάστασή μας είναι άσχημη ως προς αυτό. Ένα αίτιο είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει ότι είναι επιλέξιμη και μπορούν να πάρουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω διαφορετικών προγραμμάτων είτε εθνικών είτε απευθείας από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή η διαδικασία ενημέρωσης διαφέρει από χώρα σε χώρα στη Ρουμανία ε, έγινε μια εκστρατεία ενημερωτική το γιατί το, την περίοδο 2007-2013, αλλά ήταν σταγόνεν το ωκεανό. Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Εθνικά Κοινοβούλια και πάνω απ' όλα οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα για να ενημερώσουν τον κόσμο και να δώσουν στον κόσμο κίνητρα για να συμμετέχουν σε προγράμματα. Αυτό είναι, πιστεύω, ένα βήμα που πρέπει όλοι από κοινού να θεωρήσουμε προτεραιότητα. Και ένα δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω εδώ αφορά στις ε, δημόσιες αγορές. Το 43% σύμφωνα με μια τελευταία ανάλυση των λόγων για τι είναι τόσο χαμηλή η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων σε ορισμένες χώρες έχουν να κάνουν με τις ε, δημόσιες αγορές. Εδώ πρέπει όλοι να κάνουμε προσπάθεια και να εισαγάγουμε κάποια ελάχιστα κοινά στάνταρ για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των ενωσιακών κονδυλίων, αλλά και να βελτιώσουμε και τον αντίκτυπο που θα έχουν αυτά. Είναι αυτές δύο προτεραιότητες λοιπόν που πρέπει να μας απασχολήσουν. Ε, αναφερθήκατε βέβαια στις ε, εξάντε conditionalities, αλλά πολύ γενικά. Γι' αυτό ρωτώ συγκεκριμένα κύριε Επίτροπε εσάς. Πώς πιστεύετε ότι οι χώρες θα επιτελέσουν πρόοδο σε αυτά τα δύο θέματα και τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν και τι συνιστά η Κομισιόν να γίνει. Ο Επίτροπος Χάν και βεβαίως αν, θέλουν, αν θέλει και, ο κύριος, και οι κύριοι πρέσβοι να ε, μιλήσουν θα έχουν το λόγο. Ευχαριστώ. Θυμίζω καταρχήν ότι αλλάξαμε την πολιτική μας, δηλαδή στις τωρινές δημοσιο... προοπτικές ε, οι επενδύσεις στην υποδομή είναι στην καρδιά των επενδύσεων τώρα είναι η προώθηση της οικονομίας που δεν αποκλείει και επενδύσεις σε ε, ε, ε, υποδομές αν χρειάζεται. Στην Λετωνία για παράδειγμα έγινε πολλές φορές αυτή η συζήτηση και ένας λόγος για τη μετανάστευση είναι η χαμηλή μισθή και η δυνατότητα να κερδίζουν πολύ περισσότερα στο εξωτερικό. Για να μείνει ο κόσμος στη χώρα πρέπει να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση. Θα πρέπει να δημιουργηθούν επιχειρήσεις, να αυξηθεί η απασχόληση, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να αυξηθούν οι μισθοί, τα εισοδήματα. Αν επενδύσουμε μόνο στις υποδομές δεν θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να τα κάνουμε και τα δύο, ούτως ώστε να, να... εξελιχθούν οι χώρες αυτές ακούσαμε σχόλια από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Νομίζω ότι γι' αυτό θέλουμε να έχουμε αυτές τις έξυπνες εξειδικεύσεις και συσπυρώσεις, κλάστερς, για να μάθουμε σε κάθε περιφέρεια ποιες δυνατότητες υπάρχουν να διευρυνθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες για να διατηρηθούν και ακόμα καλύτερα να δημιουργηθούν και άλλες θέσεις εργασίας. Πάνω απ' όλα πρόκειται για την προσφορά ευκαιριών και προοπτικών ε, στους ανθρώπους της περιφέρειας όπου μένουν. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να μείνουν εκεί που ε, έχουν γεννηθεί, αλλά να έχουν και προοπτικές για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, ότι μπορούν να παραμείνουν εκεί. Αυτό πρέπει να τους προσφέρουμε. Ο, ένας συμπατριώτης μου με ρώτησε για τους δείκτες. Έχουμε δείκτες, τους χρησιμοποιούμε και μετράμε ακριβώς αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε αναφέρομαι στον τρίτο πυλώνα της πολιτικής μας να συμφωνήσουμε για ποσοτικά προσδιορίσιμα αποτελέσματα που θα φαίνονται και θα κοινοποιούνται στο τέλος της προγραμματικής περίοδου ούτως ώστε ο καθένας, κάθε πολίτης να παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών μας τι αποτέλεσμα έχουν και αν δεν έχουν αποτέλεσμα υπάρχει δυνατότητα να τεθεί θέμα να ασκηθούν ε, δημόσιες και πολιτικές πιέσεις. Δηλαδή και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο διαφάνειας που βελτιώνει ακόμα περισσότερο την αποδοχή των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τώρα, για την εξάντε conditionality, εδώ δεν πρέπει να συγχαίουμε ε, έννοιες. Οι μακροοικονομικές προϋποθέσεις και η αιρεσιμότητα ε, δεν έχει να κάνει με τους εκ των προτέρων όρους ή το εξάντε conditionality. Όταν μιλάμε για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα, αυτή έχει να κάνει με την απόδοση των κρατών μελών κατά τη διάρκεια των προοπτικών. Και για να είμαι ειλικρινής, το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι μεταξύ 50 και 95% και στην Ιταλία σε κάποιες περιφέρειες είναι 50% και ακόμα παραπάνω. Και αν η μακροοικονομική απόδοση του κράτους μέλους δεν είναι τέτοια ώστε να μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν κάτι που αποτελεί την φτηνότερη ευκαιρία για να καταπιαστούν με κάτι, πρέπει να το δούμε και να αλλάξουμε την κατάσταση και να δώσουμε στα κράτη-μέλη, στους τελικούς αποδέκτες κλπ. τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα κονδύλια. Πρέπει να παρεμβαίνουμε. Αλλά όπως ελέγχθηκε, τονίστηκε πολλές φορές και συζητήθηκε στο Κοινοβούλιο και αλλού, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα ε, είναι η τελευταία καταφυγή. Αν όλα τα άλλα έχουν εξαντληθεί, όλα τα άλλα μέτρα δηλαδή, ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη-μέλη. Δεν αρχίζουμε με την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Αυτή εφαρμόζεται με πολλούς εκκλητικούς παράγοντες και παράγοντες μετριασμού ανάλογα με την οικονομική κατάσταση ενός κράτους μέλους όταν ε, επανειλημμένα αρνούνται να λάβουν μέτρα για να βελτιώσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Για το ΑΕΠ και άλλα στατιστικά στοιχεία που ε, ζήτησε η κυρία Τέγκρα από τη Δανία. Κανείς δεν είναι ευτυχής επειδή το ΑΕΠ είναι το μόνο αποφασιστικό κριτήριο για τον υπολογισμό της κατανομής των κονδυλίων, αλλά μέχρι τώρα, κυρίως μεταξύ κρατών μελών, δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε επί πρόσθετων ε, στοιχείων. Παράδειγμα, κάποια κράτη-μέλη θα ήθελαν να λαμβάνεται υπόψη το υψηλό ποσοστό ανεργίας. Ενώ άλλες, και αυτό δεν εκπλήσει, είναι αυτοί που πληρώνουν τα περισσότερα, ε, πιστεύουν ότι μια χώρα με υψηλή ανεργία δεν πρέπει να ανταμείβεται επειδή έχει υψηλή ανεργία, παίρνοντας και άλλα λεφτά. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι σκέψη ανάλογα από τα κράτη-μέλη. Επί του παρόντος, το μόνο στοιχείο επί του οποίου μπορέσαμε να συμφωνήσουμε, τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν, είναι το ΑΕΠ. Γίνονται κάποιες συζητήσεις, γιατί κάποιοι θέλουν κι άλλα στοιχεία και άλλους δείκτες που θα απεικονίζουν καλύτερα και ακριβέστερα την κατάσταση. Τώρα όμως έχουμε το ΑΕΠ. Πάντως θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση προσθέτοντας και άλλους δείκτες. Και ένα τελευταίο σχόλιο που έθεσε ο Κροάτης συνάδελφος προς το τέλος και μου δίνει αυτό την ευκαιρία να προσθέσω κάτι ακόμα για τους ε, τερματικούς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Υπάρχει, μια, υπάρχει το νησί Καρκ. Υπάρχει και άλλη ιδέα να γίνει κάτι παρόμοιο στο Κόπερ στη Σλοβενία και δίπλα στο λιμάνι της Τεργέστης να υπάρχει κι άλλος θερματικός ε, υγροποιημένου αερίου. Για όλη την περιφέρεια όμως αρκούσε ένας θερματικός ε, LNG, υγροποιημένου φυσικού Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να βρεθεί μια συμφωνία. Πού θα γίνει τέλο πάντων ο τερματικός του LNG. Και αν μιλάμε, αν μιλάμε και για ευρωπαϊκά κονδύλια, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ε, σε μια απόσταση 100-150 χιλιόμετρων Τρει σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, δεν μπορούμε να το δώσουμε. Μπορεί κανείς να πει ένα δεν φτάνει, πρέπει να υπάρχουν διασυνδέσεις προ την ενδοχώρα και αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Αυτά ποιο θα τα πληρώσει, πώς θα γίνουν οι διασυνδέσεις και ποιε θα είναι οι διασυνδέσεις στην ενδοχώρα. Υπάρχουν πολλές ανάγκες ε, για διευκρινήσεις και επεξηγήσεις. και αυτό είναι κομμάτι της πολιτικής μας και ρωτώ, ζητώ από την Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία να συντονιστούν μεταξύ τους. Θα ήταν πολύ καλό να βρεθεί μια λύση και να μην χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίξει ρόλο διαιτητικό. Πάντως είναι σημαντικό να συζητηθεί το θέμα και να βρεθούν λύσεις και τρόποι επίλυσης ε, ξανα, να σας ευχαριστήσω για τις ε, παρεμβάσεις σας, για τον ενθουσιασμό σας που ήταν προφανής. Η ιδέα του συμπατριώτη μου για τις συμφωνίες εταιρική σχέσης που δεν πρέπει μόνο να συζητείται αλλά να υιοθετηθεί και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων ε, για να μάθουν περισσότερα πράγματα όλοι. Αυτό το κρατώ εγώ. Βέβαια ε, έχουν ήδη ε, θεσπιστεί και εγκριθεί με συγκεκριμένο τρόπο. Και τώρα ο πρέσβης κύριος Σωτηρόπουλος. Thank you, uh, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μία πολύ σύντομη παρατήρηση ε, ο Χερντόκτορ Πιρ Κούμπερ αναφέρθηκε στη χώρα μου και συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρηση που έκανε. Νομίζω ότι αναφέρθηκε στο ρόλο της πολιτικής ε, συνοχής για την ίδρυση ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτό το ανέφερε ως πολιτική συνοχής. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Thank you. So with this we finish this first... Uh, Τελειώνουμε έτσι την ε, πρώτη συνεδρία. Μισό λεπτάκι για να αλλάξουμε τις πινακίδες με τα ονόματα. Παρακαλώ πολύ μείνετε όμως στην αίθουσα. Θα ξεκινήσουμε αμέσως, αμέσως με τη δεύτερη σύνοδο. Όσοι θέλουν να παραμένουν στο δεύτερο πάνελ, στο δεύτερο τμήμα της συζήτησης, να καθίσουν παρακαλώ. Περνάμε στη δεύτερη σύνοδο. Ε, η προκλήσει σχέση με την εφαρμογή. Καταρχίζω από τον υποδιευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ρίτζιο της Επιτροπής που είναι υπεύθυνο για την ε, εφαρμογή και τον κύριο Πόπενς του ε, δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτή την πολύ σημαντική συνεδρίαση. Καλωσορίζω τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι προφανές ότι πολλά έχουν ήδη λεχθεί, δεν θα τα επαναλάβω. Να ξεκινήσω όμως εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου για το Κοινοβούλιο. Ε, που μας επέτρεψε με την ψηφοφορία να ολοκληρώσουμε τα προγραμματιστικά έγγραφα με τα κρατη να ολοκληρώσουμε εννοώ τι, τι εννοώ, ε, πρέπει να εντείνουμε την ε, διμερή, τις διμερή μας εργασίες με τα κρατη και με τις περιφέρειες, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα, έτσι ώστε τα προγράμματα, τα έγγραφα προγραμματισμού να είναι έτοιμα και να αρχίσει η η λειτουργία των ταμείων το σύντομα το δυνατό. Ο στόχος είναι βέβαια να ξεκινήσουμε το 2014, αλλά για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε πάρα πολύ στενά. Να σας ε, πω δύο λόγια το πού βρισκόμαστε, παρόλο ότι οι κανονισμοί υιοθετήθηκαν και θα δημοσιευθούν πιθανότατα λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Η Κομισιόν το ανέμενε ήδη αυτό, περιμέναμε ότι θα πάρει χρόνο. Γι' αυτό το λόγο πριν από 1,5 χρόνο προτείναμε στα κράτη-μέλη να ακολουθήσουμε μια, ε, ε, μια προσέγγιση ε, πιο βέλικτη, να ξεκινήσουμε ήδη κοιτάζοντας ποιες είναι οι ανάγκες και τα προβλήματα των κρατών και των περιφερειών και να και να ξεκινήσουμε ένα τύπο διάλογο. Συνεπώς ε, οι Υπηρεσίε κομισιών με οριζόντιο τρόπο, μια και καλύπτονται πέντε ταμεία, ε, ε, οι υπηρεσίε κομισιών συνέταξαν ένα έγγραφο για κάθε κράτος μέλος, το στείλαμε στο, στα αντίστοιχα, τα στείλαμε αυτά στα αντίστοιχα κράτη-μέλη, τους ζητήσαμε να τα εξετάσουν και να μας ενημερώσουν για τη γνώμη τους ε, σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες και τα κενά της επόμενης περίοδου 2014-2020. Τα περισσότερα κράτη-μέλη πήραν στα σοβαρά αυτό τον άτυπο διάλογο και συναντήθηκαν με τις ε, διάφορες ε, διαχειριστικές αρχές που είναι υπεύθυνε σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την προετοιμασία των προγραμμάτων. Συναντηθήκαμε ε, πολλές φορές με όλα τα κράτη-μέλη, τα μισά περίπου μας υπέβαλαν πολύ όριμες ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης ή μάλλον θα είναι έτοιμα να μας υποβάλουν επισήμως τέτοιες ε, ε, προτάσεις ε, αρχές του επόμενου χρόνου έτσι ώστε το πρώτο τρίμηνο να έχουν εγκριθεί. Παρ' όλα αυτά Όλα τα κρατημέλη έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν ένα όριμο, ε, μια όριμη πρόταση εταιρικής συμφωνίας που θα λαμβάνει υπόψη όλα όσα υπόθηκαν στην πρώτη συνεδρία. Κάθε κράτος μέλος επίσης θα πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον τρία πρόγραμμα, προγράμματα. κράτη-μέλη τα οποία επέλεξαν να έχουν περιφερειακά προγράμματα θα πρέπει να υποβάλουν μάλιστα ακόμα μεγαλύτερο αριθμό. Δηλαδή ε, θα έχουμε 28 συμφωνίες συνταρικής σχέσης και πάνω από 350 προγράμματα. Να πω 350, 500 κατά βάση αν λάβουμε υπόψη όλα τα ταμεία. Τεράστιο έργο αυτό. Ε, ας είμαστε όμως ε, έτσι λίγο ομοί. Ε, το σημαντικό είναι όλα αυτά να, έχουν, να είναι ποιοτικά και να αντικατοπτρίζουν, να πηχούν αυτά που είπαμε στην πρώτη συνεδρία σήμερα. Πού βρίσκονται τα, οι προκλήσεις. Πρώτον, η στρατηγική βάση για τις επενδύσεις του μέλλοντος. Όπως ε, είπα προηγουμένως, προσπαθούμε να απομακρυνθούμε από την λογική της απορρόφησης κονδυλίων και να προσαρμοστούμε σε μια ε, προσέγγιση επενδύσεων που θα έχουν ε, αποτελέσματα επί της ε, ανάπτυξης. Θα υποστηρίξουμε διαχρονικές μεταρρυθμίσεις και project τα οποία θα δίνουν θέση απασχόλησης και θα είναι βιώσιμα. Επίσης, καλούμε τα κράτη-μέλη να αναζητήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και τις, ε, τους τομείς στους οποίους ε, πρέπει να γίνουν επενδύσεις έτσι ώστε να α, ε, αυτών των πλέον εκτιμάτων. Ε, <clears throat> μιλήσαμε πολλές φορές για την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα και εδώ παίζει ρόλο, είναι πολύ σημαντικό τμήμα του προγραμματισμού. Η αιρεσιμότητα αυτή είναι κατά βάση οι όροι που θα πρέπει να ε, ικανοποιούνται προκειμένου να πετύχουν τα προγράμματα. Η εκ των προτέρων ερεσιμότητες ε, ορίζονται με βάση τα διδάγματα που έχουμε εξάγει και έχουμε εξαγάγει και τις σημερινές μας εμπειρίες. Υπάρχουν οριζόντιες ερεσιμότητες όπως οι μεταγραφές εθνικών οδηγιών, ε, οι, οι όροι περί δημοσιοδιαγωνισμών κλπ. Αλλά έχουμε και συγκεκριμένες ερεσιμότητες ε, ανάλογα με, τις, ε, με τους τομείς, τα master plans των μεταφορών, το, τις ευφυείς εξειδικεύσεις κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι έτοιμα πριν ξεκινήσουν οι επενδύσεις. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική χρήση των χρημάτων του φορολογούμενου και η Κομισιόν θα ε, περιορίσει ε, τις δαπάνες σε αυτούς τομείς αν δεν πληρούνται αυτές οι συνθήκες η συγκέντρωση και η απόδοση προτεραιοτήτων θα πρέπει να εξασφαλιστούν, θα πρέπει να ε, δώσουμε κάποια ευελιξία, αλλά δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε την, τον κατακαιρματισμό των κονδυλίων σε πάρα πολλούς τομείς που ενδεχομένως θα μπορούσε, να θεωρηθεί ως πολιτικά απαραίτητο, για μας όμως αυτό δεν είναι δυνατό. Θα πρέπει να συγκεντρωθούμε σε συγκεκριμένους τομείς και τα έγγραφα που έστειλε η Κομισιόν στα κρατη είναι κατά την άποψή μα πλαίσιο ε, το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη συγκέντρωση των, της προσπάθειας. Μετά, ε, θα πρέπει να προσανατολιστούμε στα αποτελέσματα. Και αυτό είναι κάτι καινούριο στο ρυθμιστικό μας πλαίσιο. Άλλαξε η όλη νοοτροπία, η λογική τη παρέμβασης. Οπότε πρέπει να δούμε τι αποτελέσματα πρέπει να επιτευχθούν Θα πρέπει οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν να είναι σαφείς, να είναι ρεαλιστικοί, να είναι φιλόδοξοι και γι' αυτό λόγο θα πρέπει να συνεργαστούμε για, τον, για την κατάρτιση των δικτών. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα από τα αδύναμα μας σημεία αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να τα καταφέρουμε πριν αρχίσουμε να ξοδεύουμε. Θα πρέπει να καθορίσουμε στόχους και δείκτες σωστά. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλους, αλλά χωρίς αυτό δεν είναι δυνατό να αποδείξουμε ότι τα καινούργια αποτελέσματα είναι αποτελεσματικά. Αλλά βέβαια όχι μόνο προγράμματα και συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Τώρα, ο στόχος είναι όλα τα έγγραφα προγραμματισμού να υιοθετηθούν μέσα στη θητεία της, ε, αυτής της Επιτροπής ε, παρ' όλα αυτά πολλά εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη και από τις περιφέρειες πόσο θα συνεργαστούν μαζί μας και πόσο γρήγορα θα μας υποβάλουν τα έγγραφα που είναι απαραίτητα έτσι ώστε να τα αναλύσουμε. Και βέβαια τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν και πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό τους επόμενους μήνες, γιατί όπως είπα οι εκ των προτέρων ερεσιμότητες ε, συνήθως απαιτούν νομοθετικές αλλαγές, τροποποίησεις, προσαρμογές, κάτι που προφανώς είναι έργο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, βέβαια, ε, επίσης υπάρχει και το θέμα του καθεσμού των προτεραιοτήτων. Η, η εταιρική σχέση έχει ήδη καταγραφεί στους κανονισμούς, αλλά τα κοινοβούλια πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο έτσι και αλλιώς για τον καθεσμό των μελλοντικών προτεραιοτήτων. Αυτά ήθελα να πω σήμερα. Είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Νόρμουντς Πόπενς. Τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, Βιργίνια Μπαλτραϊτίενε από τη Λιθουανία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ντανούτα Χιούμπνερ, την Πρόεδρο της Επιτροπής, για την πρόσκληση και όλους για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σε αυτή τη συνάντηση. Νομίζω ότι ένα ενεργός διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι αμοιβαία υποφελή άσκηση, αν θέλουμε να εφαρμόσουμε με επιτυχία τη μελλοντική πολιτική συνοχή. Θέλω να ευχαριστήσω την, Επιτροπή αυτή για την εφαρμογή αυτή τη πολιτική που είναι πολύ φιλόδοξη και ανοίγει νέε ευκαιρίε, προωθεί την ανάπτυξη, την κοινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Η σημερινή λιθουανική Προεδρία αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση. Ε, αλλά η πρόκληση αυτή αφορά όλους μας, και τους ε, υπαλλήλου και τους πολιτικούς. Πριν δύο μέρες, 25 Νοεμβρίου, ε, κάναμε στο Βίλνος μια εκδήλωση της Προεδρίας του Κοινοβουλίου και οι πρόεδροι των Επιτροπών Περιβάλλοντος, ε, των τοπικών αρχών και των Επιτροπών ε, Δημόσιας Διοίκησης συμμετείχαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τάνουτα Χιούμπνερ και τον Επίτροπο, τον κύριο Χάν, για τι καλέ παρουσιάσει και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε. Η συνθήκη Λισαβόνα αποτέλεσε τη βάση για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και στενότερου δεσμού μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του κοινού και των κοινωνιών. Ο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων έχει ενισχυθεί σημαντικά. Με το νέο ε, πολιτεύσιμο πλαίσιο, εμεί οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων μπορούμε να υποφεληθούμε πλήρως από τις ε, ευκαιρίες που έχουμε και να συμμετάσχουμε ενεργά, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την πρόοδο στις χώρες μας και στην Ευρώπη. Τα εθνικά κοινοβούλια μπορεί να γίνουν βασικοί παίχτες και εταίροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων για να διαμορφώσουν την πολιτική συνοχή και να παρακολουθήσουν την εφαρμογή τη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πλήρω τις τυπικές, επίσημες και άτυπες διαβουλεύσεις και συζητήσεις. Γίνονται συζητήσεις σε διάφορα επίπεδα, όπως ξέρετε, για τις προκλήσεις που αφορούν την πολιτική συνοχή. Και αν θέλουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά την, τα κονδύλια των διαφορετικών ταμείων την περίοδο 2014-2020, πρέπει καθώς να διδαχτούμε από τη σημερινή περίοδο προγραμματισμού που τελειώνει. Ο βασικός μας στόχος είναι να δούμε τι δουλεύει καλά και θα πρέπει να συνεχιστεί στο μέλλον, ποια ήταν τα πιο δύσκολα, δυσεπίλητα προβλήματα, τι λάθη έγιναν και τι πρέπει να αποφύγουμε βέβαια στο μέλλον. Χαίρομαι που στη Λιθουανία έχουμε ένα μοντέλο διοίκηση και ελέγχου που εξασφαλίζει υπεύθυνη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα ήθελα να σας πω ότι το κοινοβούλιο μας ήδη στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 θέτησε ένα ψήφισμα για τις κατευθυντήριες γραμμές για το Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση για να εφαρμόσει τη στρατηγική διαφορετική υποστήριξης στη σημερινή περίοδο προγραμματισμού, δηλαδή το 2007-2013. Το ψήφισμα αυτό ε, μιλάει για τις στρατηγικές προτεραιότητες προκειμένου να ενισχύσουμε την ε, οικονομία μας και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας πιο συγκεκριμένα. Κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο υποβάλλει στο συγγνώμη, η κυβέρνηση υποβάλλει στο Κοινοβούλιο ε, μία έκθεση για τις ε, τάσεις ανταγωνιστικότητας οικονομίας. Με αυτή την έκθεση ανταγωνιστικότητας λαμβάνουμε και τον πίνακα αποτελεσμάτων με τους πίνακες, με τους ε, δείκτες και κάποια κριτήρια που έχουμε προκαθορίσει, ούτως ώστε να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα προγράμματα. Με αυτό το ψήφισμα η πολιτική μας άνοιξαν ε, την εφαρμογή της, των προγραμμάτων διαρθωτικής υποστήριξης στον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Ελέγχει λοιπόν το Κοινοβουλίο και οι βουλευτές του Λιγαθιονικού Κοινοβουλίου ε, συμμετέχουν σε καθήλυνα αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για να ε, ελέγξουν τις διάφορες εκθέσεις που παρουσιάζονται ανατομέα. Ακούμε λοιπόν τις παρουσιάσεις των εκθέσεων στις διάφορες επιτροπές και νομίζω ότι αυτό ήταν αποτελεσματικό μέτρο. Ε, μας εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιοι φορείς ε, κάνουν σωστά τη δουλειά τους και οι πολιτικοί δραστηριοποιούνται έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και θα ήθελα να σας αναφέρω μερικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς, πολύ συχνά υπάρχουν ε, πολλαπλές αρμοδιότητες, δηλαδή Διάφορε επιτροπές, α πούμε η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Δημοσίας Διοίκησης και άλλες επιτροπές ε, είναι συναρμόδιες. Είναι δύσκολο όμως με αυτόν τον τρόπο να συντονιστούμε. Επίση, μερικέ φορέ δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να λάβουμε αποφάσει σε κάποιου τομεί. Επίση, έχουμε διαστάμενε απόψει όταν συζητάμε ας πούμε, ευρωπαϊκά θέματα ή εθνικά θέματα. Οι διαδικασίες της ε, πολιτικής συνοχής είναι πάρα πολύ περίπλοκες. Υπάρχουν διάφοροι φορείς, διάφοροι εξωματούχοι που συμμετέχουν και υπάρχει ένας καταιγιστικός αριθμός πληροφοριών. Χαίρομαι που αφιερώνουμε πολύ χρόνο και προσπάθεια στο, στην ανάλυση των προγραμμάτων για να δούμε τι ε, όφελο έχουν για τους πολίτες στις διάφορες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές. Και συχνά βλέπουμε ε, προγράμματα τα οποία μοιάζουν ωραία και καινοτόμα, αλλά τελικά δεν είναι αποτελεσματικά, δεν κάνουν τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εμείς οι βουλευτές θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για διάλογο, μια και αυτές είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή του προγράμματος. Δεν χρειαζόμαστε μόνο φυσικούς δείκτες, πρέπει να αξιολογήσουμε και την επίπτωση σε ένα συγκεκριμένο τομέα κοινωνικό οικονομικό κτλ. Πρέπει επίσης να ξέρουμε τις απόψεις ε, της κοινότητας, των πολιτών, ε, την αξιολόγησή τους, τις τάσεις. Νομίζω ότι με, με την πολιτική συνοχή θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε ποιοτικού δείκτες και στην παρακολούθησή τους. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε μεγάλη προσοχή στην αξιολόγηση των ε, μηχανισμών υποστήριξης και στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων και την επίπτωση που έχουν στην υλοποίηση των στόχων που έχουμε προκαθορίσει. Η μελλοντική πολιτική συνοχή έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, δείκτε εύκολη παρακολούθηση, δείκτε αξιολόγηση που εξασφαλίζουν πειθαρχία. Υπάρχουν πολλά μέτρα ίσως, αλλά αυτό που μετράει είναι το κατά πόσον υλοποιούνται οι δείκτε. Με ένα σαφέ σύστημα δικτών, το Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει το ρόλο της, ε, της επιτήρησης πολύ πιο άνετα. Και πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό. Καταρχάς ένα σαφές σύστημα παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο. Με σαφείς ευθύνε για τα διάφορα, του διάφορους φορείς και τα θεσμικά όργανα και σαφείς διαδικασίες. Οι διαδικασίες θα πρέπει επίσης να απλουστευτούν. Χρειαζόμαστε ε, σαφή ε, συστήματα και μηχανισμούς εφαρμογής. Επίσης αρμοδιότητες σαφείς για τις καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές για τα κοινοβούλια. Οι επιμέρους επιτροπές θα πρέπει να συζητήσουν για να καθοριστούν οι προτεραιότητες όσον αφορά τι επενδύσεις. Χρειαζόμαστε επίσης κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θα πρέπει να γίνεται και στις ενδιάμεσες φάσεις ενός project, ενός προγράμματος, ενός έργου. Επίσης θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα ωφέλη του προγράμματος στην ευρύτερη κοινωνία. Χρειαζόμαστε ενεργή διαβούλευση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με τα εθνικά όργανα ε, με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και με τις εθνικές κυβερνήτες. Οι απόψεις των πολιτών έχουν μεγάλη σημασία. Και φυσικά τα μέλη των ε, κοινοβουλίων εκπροσωπούν τους λαούς. Ξέρουν ε, καλύτερα τα συμφέροντά τους, τους εκπροσωπούν, εξάλλου έχουν εκλεγεί από αυτούς. Θα πρέπει η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύπτει τις ανάγκες των λαών μας. Επίσης, ε, οι τοπικές κοινότητες θα πρέπει να εμπλακούν στην ε, διαδικασία προγραμματισμού και θα πρέπει να εμπλακούμε και, στην, και εμπλακούν μάλλον στη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θα πρέπει όχι μόνο να βασιζόμαστε για την παρακολούθηση σε δείκτες και σε στατιστικά στοιχεία, θα πρέπει να υπάρχουν και δημοσκοπήσεις και σφιγμομετρήσεις. Η κοινοβουλευτική εποπτεία θα πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Η ανταλλαγή όμως καλών πρακτικών ή βέλτιστων πρακτικών, όπως η σημερινή συνάντηση, ε, άτυπες μορφές συναντήσεων, ε, αλλά και επίσημες συναντήσεις όπως η σημερινή, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Η σημερινη μπορεί να παιξουν σημαντικο εφαρμογή της πολιτικής συνοχής εξαρτάται από τη στάση μας, συμπεριφορά μας, από τη διάθεσή μας να ασχοληθούμε από το ρόλο και την ευθύνη που θα έχουν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σε ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας πω αυτές τις απόψεις για αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό και καλώ τους συναδέλφους για να πούν τις απόψεις τους. Ελπίζω να ακούσω πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις. Ευχαριστώ. Καλή τύχη. Γιάννης Κεφαλογιάννης την, Εθνική, από την Ελληνική Βουλή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ε, εκδήλωση αυτή και τη δυνατότητα που μας δίνεται να μιλήσουμε για το Ελληνικό Κοινοβούλιο ε, στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και τώρα θα μιλήσω ελληνικά. Η οικονομία είναι αποτέλεσμα παραγόντων δεκαετιών. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, χρειάζεται να συνδέσουμε άμεσα την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής με την αποκατάσταση της ανάπτυξης και ευημερίας σε κάθε ευρωπαϊκή περιφέρεια. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, το ελληνικό κατακεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης έπεσε από το 94% του μέσου κοινοτικού όρου το 2009 στο 79% το 2011, όταν το 1995 ήταν στο 84%. Δηλαδή το προϊόν της χώρας υποχώρησε σε επίπεδα της προηγούμενης 20 Το Ευρωκοινοβούλιο έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για του νέου κανόνε που θα διέπουν την πολιτική συνοχή κατά την περίοδο 2014-2020. Έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο σκληρών διαπραγματεύσεων, 325 δισεκατομμύρια ευρώ θα πάνε στι περιφέρειε τη Ευρώπη. Κυρίε και κύριοι, η ευρωπαϊκή πόρη είναι κρίσιμη για την Ελλάδα, καθώ σε μεγάλο βαθμό είναι και η κυριότερη διαθέσιμη για αναπτυξιακέ επενδύσει, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Το γεγονό αυτό καθιστά την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και την έμφαση που θα δοθεί σε αυτέ σε σχέση με τον χρόνο υλοποίηση περισσότερο αναγκαίε από ποτέ. Η αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την περίοδο 2014-2020 αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την αντιμετώπιση, στον βαθμό που τη αναλογεί, των διαθροτικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων και τη στροφή σε ένα νέο αναπτυξιακό παράδειγμα που θα είναι στηριγμένο στι δυνατότητε τη χώρα και στην εξειδίκευση και ανταγωνιστικά ε, πλεονεκτήματα των περιφερειών η βασική επιδίωξη της ελληνικής στρατηγικής για την πραγματική περίοδο 2014-2020 είναι να εξασφαλίσουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πόρων θα δράσει ως καταλήτης για την ενεργοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων την επόμενη δεκαετία. Αν επιτύχουμε σε αυτό το επιχείρημα, τότε θα εξασφαλίσουμε τις βασικές προϋποθέσεις για μια ευημερία που θα βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεών μας, εκτοστρακίζοντα την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και κάνοντας πρακτική την ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας θέμενες αξίας. Τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός και εκτός του πλαισίου 2014-2020 στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, στην επαναφορά του κατακεφαλήν εισοδήματος στα πρώτης κρίσης επίπεδα, στην αύξηση της ολικής παραγωγικότητας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών και στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων και ορατού εξυγχρονισμού του κράτους με την προώθηση του συνόλου των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τομείς. Κυρίε και κύριοι, για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της χώρας, επιλέγονται στο πλαίσιο της στρατηγικής πέντε χρηματοδοτικές προτεραιότητες που συνάδουν απόλυτα με το κείμενο θέσεων της Επιτροπής, με συγκέντρωση των πόρων σε επιλεγμένους θεματικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες Συγκεκριμένα, πρώτον, ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα και τη εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση τη εγχώρια προστιθέμενη αξία. Πρόκειται για την πιο εμβληματική. Λίγο πιο αργά να διαβάζετε αν είναι δυνατόν για να παρακολουθούν οι διερμηνείς και αυτό ισχύει για όλους. Thank you. Ε, μην μιλάτε πολύ γρήγορα. Ε, πρόκειται για την πιο εμβληματική των ε, προτεραιοτήτων, καθώς σηματοδοτεί με το περιεχόμενό της και τον ολοκληρωμένο της χαρακτήρα την κύρια στροφή στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα. Η παραγωγική, ανταγωνιστική και δυνάμει εξωστρεφή κλάδη, όπως ο τουρισμός, η γεωργία, η μεταποίηση και οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις αποκτούν κεντρικό ρόλο και σημαντικό μερίδιο στην κατανομή πόρων και επενδύσεων. Δεύτερον, ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, ενεργώς κοινωνική ενσωμάτωση. Αποτελεί επίσης μεγάλη σημασία σχηματοδοτική προτεραιότητα, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης και της ύφεσης, δηλαδή την ανεργία και τη φτώχεια. Με στοχευμένε πολιτικέ αισιοδοξούμε να αντιμετωπίσουμε τα διαρθρωτικά προβλήματα τη αγορά-εργασία. Λόγω των εκρηκτικών διαστάσεων που έχει λάβει η ανεργία, ιδιαίτερα στου νέου, άμεση προτεραιότητα αποτελούν οι δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων και των μακροχρόνια ανέργων. Μακροπρόθεσμα, ένα καλά σχεδιασμένο πλαίσιο πολιτικών και μέτρων για την αγορά εργασίας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως υποστηρικτικό εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη. Εκ πείρας αντιλαμβανόμαστε πλέον την ανάγκη για βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος την καλύτερη διασύνδεση της εκπαίδευσης, την κατάρτιση και την διαβίου μάθηση με την αγορά εργασίας, την στήριξη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και την προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά εργασίας. Ο τρίτος θεματικός στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλά επίπεδα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, παράλληλα με την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας ενεργητική αποδοτικότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί δυνητικά για τη χώρα σημαντικό πεδίο ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητα. Επόμενη, τέταρτη βασική θεματική ενότητα αποτελεί η ανάπτυξη, ο εξυγχρονισμός και η συμπλήρωση των υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος στον τομέα των μεταφορών για τη νέα προγραμματική περίοδο παραμένει η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφορών και η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών. Στις άμεσες προτεραιότητες περιλαμβάνεται επίσης η ενίσχυση της ανάπτυξης βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών σε συνέργεια με τη χρηματοδοτική προτεραιότητα προστασία του περιβάλλοντος, μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον. Στις ενεργειακές υποδομές, η εκμετάλλευση των ελληνικών εγχώριων αποθεμάτων υδρογοναθράκων αποτελεί προτεραιότητα για τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα κάψιμα. Ο εξυγχρονισμός και η επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης της ασφάλειας του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων στη διανομή ενέργειας, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά, να βελτιωθούν και να εμπλουτιστούν οι σχετικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι τοπικοί ενεργειακοί πόροι αποτελούν βασικές προτεραιότητες στον τομέα. Τέλος, βασική προτεραιότητα χρηματοδοτική για την Ελληνική Βουλή εντός και εκτός του πλαισίου του ΣΕΣ 2014-2020 αποτελεί η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υψής της σημασίας θεωρούνται όλες οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα στήριξης στου τομείς της δημιουργίας ενός φιλικού προς επιχειρήσεις περιβάλλοντος, στη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και στην αναβάθμιση των μηχανισμών σχεδιασμού, διαχείρισης, υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Κύριε και κύριοι, κρίσιμο παράγοντα για την εφαρμογή στην πράξη όλων των ανωτέρων αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, όπως έχει δείξει και μέχρι τώρα εμπειρία, η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η εμπέδωση και κυριότητα του κοινού οράματος και των επιμέρους προτεραιοτήτων. Αν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις υπό το πρίσμα μόνο των εθνικών μας συμφερόντων, κινδυνεύουμε να χάσουμε την προστιθέμενη αξία που έχει η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναπτυχθούν συνέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα εστιάζουν σε νέους κινητήρες για την ανάπτυξη, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας. Η πολιτική συνοχή είναι η κύρια πηγή των ευρωπαϊκών δημόσιων επενδύσεων για τους σκοπούς αυτούς. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα επίση να επισημάνω ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε πλέον και το επίπεδο της μακροπεριφέρειας, καθώς μια, μια μακροπεριφερειακή στρατηγική θα μπορούσε να βοηθήσει την καταπολέμηση κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ένωσης, ενισχύοντας παράλληλα την διακρατική συνεργασία και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επίτευξη της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Μέσα σε αυτό το πλέγμα καλωσορίζουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής να καταρτήσει γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα προς μια μακροπεριφερειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στη Μεσόγειο. Πέρα των όποιων διακρατικών συμφωνιών που πλαισιώνουν την οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη συνεργασία των Ευρωπαίων πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμβάλει τα μέγιστα όχι μόνο για την ανάδειξη αυτής της πραγματικότητας, αλλά και την προάσπιση της ευημερία των Ευρωπαίων μέσα από τους μηχανισμούς της Ένωσης με δικές του πρωτοβουλίες. Προσωπικά πιστεύω ότι όσο βελτιώνουμε την επικοινωνία και διευρύνουμε τη θεσμική συνεργασία ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο τα πρώτα αντιλαμβάνονται συνολικότερα τα εθνικά του θέματα, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο αποκτά σε σχεδόν πραγματικό χρόνο καλύτερη γνώση των προκλήσεων και των προβλημάτων της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Το τελευταίο δε θα προσδώσει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στην διαχείριση κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ταχεία αντιμετώπιση τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στο μόνιμο μέλος αυτών των συνεδριάσεων που εκπροσωπεί και τον Bundesrat, την Άνω Βουλή της Γερμανίας και την Σαξονία Άνχαλτ. Ε, να μην διαβάζετε ή μιλάτε πολύ γρήγορα για τους διερμηνείς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ε, ευρωπαϊκή ε, θεσμοί ε, αναφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο και τα ταμεία παίζουν ρόλο για την υποστήριξη μέτρων, για την στρατηγική, υποστήριξη της στρατηγικής 2020 στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Ε, υπάρχουν ε, ε, σχέδια για μεταρρυθμίσεις και συστάσεις για τα κράτη-μέλη τα διαρθωτικά ταμεία, τα επενδυτικά ταμεία δεν είναι ταμεία ε, που μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε, αλλά ε, μπορούν και πρέπει με τον ιδιαίτερο τρόπο τους να συμβάλλουν στη συνοχή και την επίτευξη των βασικών στόχων της Ευρωπα... Ευρώπης 2020. Όσο περισσότερο ασχολούμεθα με την κατάρτιση συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών σχεδίων, τόσο περισσότερο νιώθουμε τις εντάσεις, το πεδίο τάσης που υπάρχει μεταξύ των στόχων Ευρώπη 2020 και των περιφερειακών και τοπικών αναγκών, αναπτυξιακών αναγκών. Τώρα, πώς μπορούμε αυτό το πεδίο τάσης να το αξιοποιήσουμε θετικά, ούτως ώστε να μην οδηγεί σε αντιφάσεις και την ε, ε, να μην, ώστε να, να μην έχουμε αποτυχίες στους στόχους της Ευρώπης 2020. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την εδαφική διάσταση. Πρώτα πρέπει να την ορίσουμε τη διάσταση αυτή πολύ καθαρά για να μην καταλαβαίνουμε διαφορετικά πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω μια τρισδιάστατη αντίληψη ή μοντέλο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εξίσου από το ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο. Η πρώτη διάσταση αυτή της εδαφικής ισορροπίας αποσκοπεί στην επίτευξη ισορροπίας οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων διαφορετικών περιφερειών μέσα από τη διαρθρωτική προώθηση και ανάπτυξη του ενδογενούς περιφερειακού δυναμικού τους. Η δεύτερη διάσταση της ε, ε, δαφικής ε, ολοκλήρωσης, υποχρεώνει τους πολιτικούς παράγοντες στην Ευρώπη να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους με τρόπο συνεκτικό, οριζόντιο και κάθετο και η τρίτη διάσταση της περιφερειακής διακυβέρνησης απαιτεί δικτύωση των δημοσίων ιδιωτικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών. Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 με τους ε, βασικούς στόχους ε, και τη μεθοδολογία καθοδήγησης μας δίνει ένα μέσον ούτω ώστε να συνδυάσουμε ευρωπαϊκούς στόχους με εθνικές, περιφερειακές και κοινοτικές ανάγκες ανάπτυξης. Ε, παράλληλα με τον κοινό προσανατολισμό έχουμε και ένα επαρκές περιθώριο για ευέλικτες λύσεις έξυπνες και καινοτόμες για τα προβλήματα επιτόπου. Ανάλογα με τα ειδικά προβλήματα, τα κράτη και οι περιφέρειες μπορούν να διαχειριστούν διαφορετικά τους στόχους Ευρώπη 2020. Για τα κράτη-μέλη τα ίδια αυτή η διαδικασία ε, διαρθρώνεται μέσα από τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τις ε, εθνικές συστάσεις. Για τις περιφέρειες ε, έχουμε τα προγραμματικά σχέδια, τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης, τα επιχειρησιακά προγράμματα. Αυτά είναι ο βασικός μοχλός για τον προσανατολισμό των αναπτυξιακών στρατηγικών επιτόπου προς την Ευρώπη 2020. Αν και δεν υπησέρχεται σε περιφερειακές διαφοροποίησεις, η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να εφαρμοστεί στις ευρωπαϊκές περιφέρειες με τις ειδικέ τους ανάγκες προκειμένου να έχει επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι οι επιμέρους περιφέρειες, ανάλογα με τα περιφερειακά τους χαρακτηριστικά, ε, με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικό βαθμό μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των εκάστοτε εθνικών τιμών στόχο. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι εθνικές τιμές στόχοι δεν μπορούν να ισχύουν σε όλες τις περιφέρειες. Πρώτον, υπάρχει πολλές φορές μεγάλη απόσταση από την πραγματική κατάσταση προς την επιθυμητή. Σε ορισμένες περιφέρειες ή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες μπορεί να μην είναι ε, ούτε ευκταίο ούτε επιθυμητό όλες οι περιφέρειες να επιτύχουν τους ίδιους στόχους. Τέλος υπάρχουν πολύ διαφορετικές δυνατότητε και δυναμικές ανάλογα για το πώς οι επιμέρους περιφέρειες συμβάλλουν στους στόχους. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της εδαφικής συνοχής θα πρέπει να δούμε πώς χωρίς σχηματικές προδιαγραφές εθνικών ε, τιμών στόχου μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι πρώτον οι πιο αδύναμες περιφέρειες δεν θα υπολείπονται ακόμη περισσότερο και θα αποσυνδεθούν από την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και πόσοι οι ισχυρότερες περιφέρειες μπορούν να συμβάλλουν στην Ευρώπη 2020 ούτως ώστε συνολικά η Ευρώπη να επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχους. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 υπ' αυτή την έννοια έχει, ενέχει τον κίνδυνο κάποιας περιφερειακής πόλωσης. Αναφέρθηκε αυτό σε ένα βαθμό σήμερα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την προγραμματική περίοδο θα πρέπει να αναπτύξουμε σενάρια που θα λαμβάνουν υπόψη τις επιμέρους ανάγκες ε, και θα τις φέρνουν σε εναρμόνιση με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Ε, εδώ υπάρχουν τέσσερα σενάρια. Το πρώτο σενάριο ε, στηρίζεται στη σκέψη ότι οι πιο σημαντικές περιφέρειες μπορούν περισσότερο να κάνουν περισσότερες προσπάθειες και να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Εδώ οι πιο ισχυρές περιφέρειες θα είναι οι ατμομηχανές για την επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων. Το πρόβλημα όμως είναι ότι με αυτό το σενάριο οι περιφερειακές ανισότητες μπορεί να επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο. Το δεύτερο σενάριο στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι πιο αδύναμες περιφέρειες σε σχέση με το σημείο εκκινήσεώς τους μπορούν να συνεισφέρουν με παρόμοιο τρόπο. Ε, έτσι όμως ε, δεν μειώνονται οι περιφερειακές ανισότητες, παραμένουν ε, αμετάβλητες. Το τρίτο σενάριο είναι το αντίθετο του πρώτου. Στηρίζεται στην υπόθεση ότι για τις ισχυρότερες περιφέρειες ε, δεν υποθέτουμε πάντα ότι την προσφορά τους θα μπορούν να την κλιμακώσουν ακόμα περισσότερο, να την μεγαλώσουν. Εδώ το μεγαλύτερο δυναμικό είναι στις πιο αδύναμες περιφέρειες που θα ανακάμψουν και θα συμβάλλουν περισσότερο στην επίτευξη των στόχων του 2020. Ε, με αυτό το σενάριο μπορούν να μειωθούν περισσότερο οι εδαφικές ανισότητες, οι στόχοι του Ευρω... της Ευρώπης 2020 και οι στόχοι συνοχής εδώ συνδυάζονται με τον καλύτερο τρόπο. Τέλος, κανένα από αυτά τα σενάρια δεν θα ε, ισχύει με τον ίδιο τρόπο για όλους τους τομείς της πολιτικής. Κάθε περιφέρεια με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο θα συμβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Σχηματοποιημένες συνταγές δεν βοηθούν πολύ. Στην τρέχουσα προγραμματική διαδικασία σημαντικό θα είναι να επεξεργαστούμε ε, τον, την αναπτυξιακή οδό που ταιριάζει στην κάθε περιφέρεια και αυτό δεν έχει σχέση με αφαίρετες επιλογές. Για να ενισχύσουμε την ε, εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής χρειάζεται η μέγιστη δυνατή ευελιξία κατά την εφαρμογή των νέων κανονισμών για τα ταμεία. Αναμφίβολα η Στρατηγική Ευρώπη 2020 ενδείκνυται ε, για να συντονίσει ε, τομεακές στρατηγικές, να βελτιώσει την εδαφική τους ε, επίπτωση, τον αντίκτυπο που έχει και να αποφύγει αρνητικές επιπτώσεις αντιτιθέμενων μέτρων. Ε, μια ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη θα επιτύχει βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ε, αηφορίας, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής. Στην ε, τρέχουσα προγραμματική περίοδο αυτή η προσέγγιση όμως δεν πρέπει να συγχαίεται με τη συγκέντρωση των προδιαγραφών και τη το μονόπλευρο προσανατολισμό της πολιτικής συνοχής ε, σε, ε, στις πανευρωπαϊκές επιπτώσεις της. κάποια παραδείγματα εδώ. Οι νέοι κανονισμοί για τα ταμεία πολύ σωστά προβλέπουν υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, ούτως ώστε η μόχλευση των κονδυλίων να αυξηθεί. Έχει νόημα όμως για συγκεκριμένες περιφέρειες ε, να περιορίζομαι τη συγκέντρωση των θεματικών στόχων εκ των προτέρων σε τρεις, αν οι ε, κανονισμοί επιτρέπουν και τέσσερις θεματικούς στόχους. Καταρχήν δεν έχουμε καμία αντίρρηση στις λεγόμενες κριτικές μάζες, αν θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε την ε, αποτελεσματικότητα των κονδυλίων. Αν θέλουμε όμως να το πάμε λίγο στα άκρα αυτό το επιχείρημα, συρρυκνώνεται στην αόριστη πίστη ότι το πολύ βοηθάει πολύ που δεν λέει και πολλά. Ε, βέβαια, εγώ την προσέγγιση αυτή του ολοκληρωμένου προγραμματικού σχεδιασμού το αντιλαμβανόμουν διαφορετικά, μάλλον σαν συνταγή μαγειρικής. Το γλυκό στον, στο μενού που ακούσαμε μπορεί κατά 80% να αποτελείται από τρία συστατικά, αλεύρι, βούτυρο, ζάχαρη. Αλλά αν λείψουν ε, τα καρικεύματα που μπορεί να μην έχουν ε, μεγάλο ποσοστό στο όλο το γλυκό, μπορεί να είναι 1%, τότε μπορεί να είναι άνοστο το γλυκό ή και πολύ ε, δυσάρεστο. Αυτά τα μικρά συστατικά λοιπόν έχουν τη μεγαλύτερη μόχλευση πολλές φορές. Οπότε έχει νόημα ε, αν έχουμε επιτύχει ένα βαθμό συγκέντρωσης 80% για το υπόλοιπο 20% να προβούμε σε περιοριστικά μέτρα, ούτω ώστε για παράδειγμα ε, τα, να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για ανταλλαγή ε, εμπειριών και για την ευρωπαϊκή δικτύωση των διοικητικών ε, επιπέδων παρόλο που η κοινωνικο-οικονομική ανάλυση εδώ δείχνει κάποιες αδυναμίες. Ε, αν λάβουμε υπόψη μας επαρκώς την περιφερειακή διάσταση και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της αναλύσεις περί αναγκών ε, τη στηρίξει ε, σε επίπεδο κράτους μέλους, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις, το περιφερειακό επίπεδο και, όπως στα, στα ευρυζωνικά δίκτυα, η πολιτική συνοχή ε, θεωρώ ότι θα έχανε το σημείο κίνησής της ε, κατά την ανάπτυξη του ενδογενούς δυναμικού στην περιφέρεια ε, αν δεν είχε τη δυνατότητα στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες επιμέρων περιφερειών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να συνδέσουμε την πολιτική 2020 ε, με μια νέα πολιτική συνοχής, ιδιαίτερα να θέσουμε ε, σημαντικές, ε, υψηλές προϋποθέσεις στην, από την, και να, να, να ζητήσουμε να λαμβάνει την υπόψη η περιφερειακή διάσταση και ο περιφερειακός αντίκτυπος. Χρειάζεται πάνω απ' όλα να υπάρχουν λύσεις ευέλικτες και όχι συγκεντρωτικές προδιαγραφές. Οι υπεύθυνοι για τη νέα πολιτική συνοχή θα πρέπει από κοινού με τρόπο συνεκτικό και διατομεακό να αναλάβουν ο καθένας τις ευθύνες τους. Ε, ε γι' αυτό χρειάζεται αμοιβαία σχέση, σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλή συντονιστική μηχανισμή που τους διαθέτουμε. Τέλος, ε, η περιφερειακή διακυβέρνηση, το governance, ε, μας δίνει τη δυνατότητα να ε, συνδυάσουμε ε, δημόσιους, ιδιωτικούς ε, παράγοντες, παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, ούτως ώστε να αναδείξουμε τη χρησιμότητά τους. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη διάμεση αξιολόγηση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, χρειάζεται την περιφερειακή διάσταση, αυτήν την place-based approach όπως τη λέμε, να την ενισχύσουμε με συνέπεια. Χαίρομαι διότι η Επιτροπή των Περιφερειών ε, ασχολείται επίσης πάρα πολύ ε, στα πλαίσια του νέου προσανατολισμού της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Νομίζω ότι ε, αυξάνονται οι αμοιβαίες σχέσεις, η παγκόσμια δικτύωση Άρα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία για την ε, αηφόρο ανάπτυξη και καλή ποιότητα ζωής για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό χρειάζεται να βρούμε μια νέα ισορροπία μεταξύ της ε, κεντρικής ε, καθοδήγησης και της αποκέντρωσης του παγκόσμιου στοιχείου, του τοπικού στοιχείου, της συναπόφασης και συμμετοχής των πολιτών και της ε, εμπλοκής των εμπειρογνωμόνων. Αυτό χρειάζεται ακριβώς, ούτως ώστε να ενισχύσουμε την περιφερειακή διάσταση της νέας πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ πολύ. Ε, περνάμε στο κυβερνοβούλιο της Δανίας, η κυρία Ντέγκερ. Ε, μιλάμε για... Έχουμε μιλήσει πολύ για βιωσιμότητα, για διατρισιμότητα σήμερα. Αν μια ευάλωτη τοπική κοινότητα γίνει πιο βιώσιμη, ε, μάλλον για να γίνει πιο βιώσιμη, θα πρέπει να ε, δούμε πώς αντιμετωπίζουν την έννοια της βιωσιμότητας οι ίδιοι καταναλωτές. Να σας πω πώς οι Δανέζοι καταναλωτές την αντιμετωπίζουν. Η αγάπη η ειρήνη και η κατανόηση <laughs> δεν λειτουργεί για να γίνει ο κόσμος καλύτερος κατά τους δάνους καταναλωτέ. Αυτό που μετράει για αυτούς είναι οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, ο χώρος εργασίας τους και η τοπική κοινότητα στην οποία ζούνε. Ανησυχούν για την κοινότητά τους, ανησυχούν για το περιβάλλον τους. Συνεπώς, αν θέλουμε να αλλάξουμε την ε, βιωσιμότητα και την έννοια της, θα πρέπει να δούμε πιο κοντά στους ανθρώπους και όχι πιο μακριά. Απ' την άλλη μεριά, οι καταναλωτές ε, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι πιο ακριβά αν αυτό διατηρεί τις θέσεις στην κοινότητά τους. Τους αρέσει η κοινωνική πτυχή των πραγμάτων, τους αρέσει να αισθάνονται τμήμα ενός ε, πιο ε, ευρέως συνόλου. Τους ενδιαφέρει να αισθάνονται καλύτερα με τις οικογένειές τους, με τους γείτονες, με την κοινότητά τους. Και επίσης τους αρέσει πολύ να αποταμιεύουν. Δεν τους νοιάζει να Παίρνουν κάποιους μικρούς κινδύνους, αλλά όχι πολλούς ούτε πολύ μεγάλους. Και τέλος, οι καταναλωτέ θέλουν να γνωρίζουν τι έχουν να κερδίσουν οι ίδιοι από οποιαδήποτε θυσία κάνουν. Θέλουν την αλλαγή σε τοπικό επίπεδο, τους ενδιαφέρει περισσότερο η οικογένειά τους και η κοινότητά τους, τους ενδιαφέρει να αισθάνονται τμήματα ενός συνόλου, δεν θέλουν να παίρνουν πολλά, πολλά ρίσκα και δεν θέλουν να πληρώνουν και πάρα πολύ. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη γνώση έτσι ώστε να κάνουμε απο, ε, παραγωγικές και βιώσιμες επενδύσεις στη Δανία. Να σας πω, στη Δανία έχουμε ένα πολύ ωραίο νησί, το Samsung, όπου ζουν περίπου 4.000 άτομα. Ε, αυτό το νησί έχει τα γνωστά προβλήματα, πολλά από τα γνωστά προβλήματα των ε, περιφερειακών περιοχών, ε, αστιφιλία, εγκατάλειψη κλπ. Ε, είπαν λοιπόν ε, ότι ε, κάποια στιγμή δεκαετία του 90 ότι σε 10 χρόνια το νησί θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα, πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο ε, πώς θα μπορούσαν όλοι να συμμετάσχουν σε αυτό το στόχο ε, με τη συμμετοχή. Όχι όμως όπως λένε συνήθως οι πολιτικοί να ε, συμπεριλάβουμε τους πολίτες μας να συμμετάσχουν κλπ. Όχι με λόγια, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πώς έγινε με το να πάρουμε σοβαρά υπόψη τη γνώμη αυτών των κατοίκων. Είπαμε, 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους ρωτήσαμε τι πρέπει να κάνουμε. Ε, κάποιοι είπαν ε, εγώ θέλω από τα άχυρά μου, γιατί είμαι γερός, θέλω τα άχυρά μου να πάρω βιομάζα. Κάποιος άλλος είπε να αγοράσουμε ανεμογεννήτριες. Κάποιος άλλος ε, είπε να εξασφαλίσουμε ένα σύστημα τηλεθέρμανσης. Οπότε κάναμε όλα όσα μας ζήτησαν. Ε, κάποιοι αγοράζουν την βιομάζα του Γεωργού, οπότε αυτός μπορεί να μείνει εκεί που είναι για να μην χρειάζεται μεταναστεύσει. Κάτι πλήρωσαν όλοι, κερδίζουν όμως πάρα πολλά και ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν κιόλα. Και δουλεύουν και πιο πολύ. Όλοι αναρωτιόντουσαν τι έχουν να κερδίσουν. Ε, ο Γεωργός βρήκε πολύ καλή ιδέα να κάνει το αχυρό του ε, ενέργεια αλλά ο ξενοδόχος ε, ε, νοικιάζει τα δωμάτια του σε πάρα πολλούς άνθρωπους που έρχονται από όλο τον κόσμο για να δουν ε, τα αποτελέσματα αυτού του project. Πολλές θέσεις εργασία δημιουργήθηκαν σε μια μικρή κοινότητα σε ένα νησί το οποίο πραγματικά είχε πληγεί από την αστιφιλία. Όλοι αυτοί ήταν τμήμα ενός ευρύτερου project. Η ανανεώσιμη ενέργεια ήταν το αντικείμενο αυτού του σχεδίου οι... εγκαταστάθηκαν ανεμογεννήτρε. Θυμάστε, ξέρετε τι γίνεται όταν εγκαθιστούμε και ανεμογεννήτρε κοντά σε κοινότητε. Ε, ε όλοι αρχίζουν και λένε «Α, είναι πολύ μεγάλο, κάνει θόρυβο κλπ. κλπ». Αν όμω εσύ είσαι ο ιδιοκτήτη αυτή τη ανεμογεννήτρια, αν ξέρει ότι η ενέργεια που θα παράξει θα είναι 100% οικολογική και θα τον αφορά γιατί θα είναι ενέργεια για τον ίδιο και για το σπίτι του, τότε αυτός ο άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι λένε «Χα, λέει, αυτή είναι η δική μου ανεμογεννήτρια και είναι όμορφη». Όλοι θεωρούν ότι οι ανεμογεννήτρες είναι πιο όμορφες επειδή ακριβώς είναι δική τους περιουσία. Είναι δικό τους περιουσιακό στοιχείο και παράγει ενέργεια για τους ίδιους. Ε, και τώρα πρόκειψε μια καινούρια φιλοδοξία. Μέχρι το 2030 δεν θέλουν να χρησιμοποιούν καθόλου ε, ορυκτούς υδρογονάνθρακες πλέον στο νησί. Έτσι κι αλλιώς τα δύο τρίτα των ε, κρατικών αυτοκίνητων στο νησί είναι ηλεκτρικά. Ε, κινούνται με ε, ηλιακή ενέργεια. Παλιότερα το νησί ήταν προβληματικό. Κλείνανε επιχειρήσει, αυξανόταν η ενέργεια. Τώρα είναι πρότυπο χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οπότε πρέπει να βασιστούμε στα ε, στους πόρους που έχουμε αντί να εισάγουμε. Βέβαια, ε, στον ε, παγκοσμιοποιημένο κόσμο η κατανάλωση αφορά αγαθά τα οποία έρχονται από όλο τον κόσμο και είναι δύσκολο να το πεις αυτό που λέω αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτα να εκμεταλλευόμαστε τους δικούς μας πόρους, τα δικά μας ατού ιδιαίτερα για, τις, για τη μικρομεσαία τάξη ε, και οι πολιτικοί θα πρέπει να βασιστούν σε αυτό και να το αναπτύξουν. Λοιπόν, και τι πρέπει να γίνει. Πρώτον, με τους κανόνες θα πρέπει να είμαστε λιγότερο γραφειοκρατικοί. Την πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου εμείς καθορίζουμε συγκεκριμένα έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν οι γεωργοί, αν θέλουν να λάβουν επιδοτήσεις κλπ. Δεν ξέρω τι γίνεται στη δική σας χώρα, αλλά στη Ιδανία... αυτοί που ζουν στην επαρχία δεν έχουν τις ίδιες, ε, τον ίδιο αλφαβητισμό ούτε τις ίδιες, την ίδια εκπαίδευση ε, που έχουν οι άνθρωποι στις πόλεις. Οπότε όταν του ε, δώσετε κάποιον ανθρώπου ένα έντυπο πολυσέλιδο δεν μπορεί καν να το συμπληρώσει. Αυτό όπως καταλαβαίνετε παρεμποδίζει την απορρόφηση των επιδοτήσεων. Μετά είμαστε διαφορετικοί. Από χώρα σε χώρα η κατάσταση είναι διαφορετική. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολο να διαθέτουμε σε ευρωπαϊκό πεδίο κανόνες που να είναι οι ίδιοι για όλους. Όταν λοιπόν έχουμε ως μοναδικό κριτήριο το ΑΕΠ, αυτό θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Όταν δούμε για παράδειγμα τις ε, αεροκατοικημένες περιοχές, τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, μας λένε δεν θέλουμε πολλά λεφτά, δεν θέλουμε κάποιος να μας στείλει πολλά κονδύλια. Εμείς είμαστε περήφανοι, θέλουμε να τα κάνουμε με δικά μας μέσα, αλλά παρακαλούμε πολύ τουλάχιστον μην μας δημιουργείτε εμπόδια. Αν πρέπει να κάνετε κάτι, αυτό δεν είναι να μας δώσετε λεφτά, να μην μας δημιουργείτε εμπόδια. Αυτό μας λένε. Και εμείς πολιτικοί αυτό πρέπει να κάνουμε. Ασφαλώς και χρειάζεται μια διαδικασία υποβολής, ε, αιτήσεων κλπ. Αλλά μην πνίγουμε με τη γραφειοκρατία ε, τις τοπικές πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ. Uh, Έχουμε 7 ομιλητέ, 3 από Εθνικά Κοινοβούλια και 4 ευρωβουλευτέ. Θα ξεκινήσω με τον Νίκο Χρυσόγελο. Πρώτος είναι αυτός ο οποίος θα μιλήσει. ο Νίκος Χρυσόγελο θα μιλήσει πρώτος. Thanks a lot. I will σας μιλήσω ελληνικά. Ε, είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων ή και Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωκοινοβουλίου. Ε, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντική γιατί μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις αλλά κυρίως και να υπάρχει μια συνεργασία πάνω σε πολιτικές που συζητιώνται. Υπάρχουν όμως πολλές πολιτικές οι οποίες σήμερα πηγάζουν κυρίως από κυβερνήσεις αλλά στην κοινωνία των, στις χώρες μας αποδίδονται σε ευρωπαϊκές πολιτικές. Μερικά παραδείγματα θα ήθελα να τα συζητήσουμε γιατί αφορά και την Επιτροπή μας εδώ. Ως Ευρωκοινοβούλιο επιδιώξαμε πάρα πολύ να υπάρχει διάλογος για την επόμενη προγραμματική περίοδο μεταξύ των κυβερνήσεων, των περιφερειών και της κοινωνίας των πολιτών για να προετοιμαστούν οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης είδαμε πολύ συχνά ότι οι κυβερνήσεις αντιδρούν πάρα πολύ στο να υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις μεταξύ αυτών τριών επιπέδων, δηλαδή κοινωνία πολιτών, περιφέρειες και κυβερνήσεις, και αρνιόντουσαν επανειλημμένα και τις δεσμεύσεις μέσα από contract, μέσα από συμβόλαια ή έστω και την πολύ πιο ήπια διατύπωση της συμφωνίας. Εκεί να χρειαζόταν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων έτσι ώστε πράγματι σε κάθε χώρα και όχι απλώς στις χώρες που έχουν παράδοση να επιτευχθεί μια τέτοια εταιρική σχέση μεταξύ κοινωνίας πολιτών, περιφερειών και κρατών ώστε μία πρώτου του 2014 να είναι έτοιμες όλες οι χώρες με ποιοτικά προγράμματα να υπογράψουν τις σχέσεις εταιρικής Τη συμφωνία εταιρική σχέση με την Κομισιόν. Ελάχιστες κοινωνίες είναι ενημερωμένε για αυτή τη δυσκολία να υπάρχει πραγματικά συμμετοχικός περιφερειακός σχεδιασμό. Το δεύτερο σε σχέση με την ε, λεγόμενη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Εδώ στο Κοινοβούλιο μεγάλη πλειοψηφία αντιτίθονταν στο να μπουν όροι όταν αποτυγχάνει μια κυβέρνηση να πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους να τιμωρούνται οι περιφέρειες και οι κοινωνίες με μείωση ή με διακοπή των χρηματοδοτήσεων, μέρους ή συνολικά των προγραμμάτων. Και 28 κυβερνήσεις, χωρίς αντίδραση από τα κοινοβούλια, υιοθέτησαν τις αρχές μακροοικονομικής αιρεσιμότητας ως όρο μέσα στους κανονισμούς των διαφορετικών ταμείων και αυτό σημαίνει ότι αύριο θα αποδίδεται στην Ευρώπη η όποια εφαρμογή της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο κατά μας υπέκυψε λάθος, αλλά δεν ψήφισε ποτέ ως Ολομέλεια, την αρχή της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Θα, προσωπικά θα περιμένω, θα προτείνω στα Εθνικά Κοινοβούλια να συζητήσουν πολύ σοβαρά τις ευθύνες των κυβερνήσεων γιατί οι πολίτες θα μεταφέρουν το βάρος στο ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε αυτόν που ήταν υπεύθυνο. Όλοι οι συγητές που προσπάθησαν να πείσουν τους ευρωβουλευτές να αποδεχτούν τη μακροοικονομική ρεσιμότητα έφεραν ως επιχείρημα ότι και 28 χώρες θέλουν να εφαρμοστεί μια τέτοια διάταξη καταστροφική για πολλούς λόγους. Το έχουμε στήσει στην Επιτροπή μας, αλλά θέλω να το ε, αναλύσω. Επίσης ένα τρίτο στοιχείο είναι το στοιχείο του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας αλλά και άλλες επιτροπές και όλα Ολομέλεια ζητούσαν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Όχι ένα άθροισμα 28 εθνικών προϋπολογισμών. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη συζήτηση μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου γιατί είναι διαφορετικό πράγμα να συζητάμε για 28 διαφορετικούς προϋπολογισμούς και διαφορετικό πράγμα να βλέπουμε τις ανάγκες μας, είτε αυτές αφορούν την καινοτομία, είτε την απασχόληση των νέων, είτε ε, τα θέματα της κοινωνικής συνοχής, είτε τα θέματα ακόμα και της ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με ευρωπαϊκούς όρους. Όχι απλώς τι θα δώσει, τι θα πάρει κάθε κυβέρνηση, αλλά πώς θα πετύχουμε ευρωπαϊκούς στόχους. Και νομίζω εκεί πρέπει να αναπτύξουμε μεγαλύτερο διάλογο. Και τέλος, ε, κλείνω με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ίσως ελάχιστα κοινοβούλια γνωρίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές έχει ασκήσει κριτική για το θέμα της προώθησης των πολιτικών της Τρόικα που είναι εκτός της λεγόμενης μεθόδου της κοινοτική, δηλαδή συναπόφαση Ευρωκοινοβουλίου, Κομισιών και Συμβουλίου. Η Τρόικα είναι ένας θεσμός ad hoc που αφασίζει χωρίς να παίρνει υπόψη ή να ψηφίζονται οι προτάσεις της ή και τα άτομά της από το Ευρωκοινοβούλιο ή να συμμετέχει το Ευρωκοινοβούλιο στην απόφαση. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές αποφάσεις του Κοινοβουλίου και μάλιστα προκάλεσε και μια δικασία λογοδοσία της Τρόικα μετά από πρόταση της δικιάς μας ομάδας. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό νομίζω για όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η έκθεση που ήταν και εξαπλό πακέτο έλεγε και λέει το Κοινοβούλιο όταν μια πολιτική δεν επιτυγχάνει τους μακροοικονομικούς στόχους, έχει παράπλευρες απώλειες, αυτή η πολιτική πρέπει να διορθώνεται και να, να υπάρχει διάλογος όχι μόνο με την κυβέρνηση του κράτους μέλους, αλλά με την κοινωνία των πολιτών. Και δύο βασικά στοιχεία είναι ότι δεν πρέπει να πλήττει η δημοσιονομική πολιτική την υγεία, την παιδεία και επίση τον κοινωνικό διάλογο. Δηλαδή δεν πρέπει να επιβάλλονται με νομοθετικέ ρυθμίσει θέματα που είναι αντικείμενο του κοινωνικού διαλόγου. Δεν ξέρω πόσα εθνικά κοινοβούλια γνωρίζουν αυτή την απόφαση, αλλά δεν έχει πραγματικά υπάρξει η αντίστοιχη συνεργασία μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων πάνω σε κάτι το οποίο είναι καθοριστικό και θα καθορίσει νομίζω και το μέλλον των ευρωεκλογών. Πάντως το Ευρωκοινοβούλιο έχει ξεκινήσει κοινοβουλευτικές επιτροπές, ελπίζω και η δικιά μας Επιτροπή αύριο και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, να συζητήσουν αυτά τα θέματα και να ξεκινήσει η λογοδοσία, να δούμε τι πέτυχε και τι είχε αποτύχει στις πολιτικές Τρόικα και θα συνταχθεί έκθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα κατεθεί στους προέδρους των πολιτικών ομάδων τον Απρίλιο. Θα ήταν καλό στα κοινοβούλια των χωρών της κρίσης μια ειλικρινής συζήτηση σε βάθο, όχι μια αψημαχία, να ξεκινήσει και να καταλήξει συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε και άλλες κρίσεις στο μέλλον, όχι με τον τρόπο που έγινε η αντιμετώπιση κρίσης τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Ο κ. Αντώνιο Λάργο Δενάντες από την Ισπανική Γερουσία. Η επιτροπή αυτή κατά την άποψή μου είναι επιτροπή σφαιρική το στην πρώτη συνεδρία συζητούσαμε τι είναι η κοινωνική οικονομία, ε, τι είναι οι ε, ε, περιοχές και τι σημαίνει συνοχή εκεί πέρα. Δεν μου απάντησε ο Πίτροπος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Χαίρομαι που εγκρίθηκε ένας προϋπολογισμός και ελπίζουμε ότι στον οδικό χάρτη υλοποίηση του ε, προϋπολογισμού με ευρωπαϊκή συνοχή θα αξιολογηθεί το κατά πόση συνοχή περιέχει αυτός ο προϋπολογισμός. Και δύο ακόμα σχόλια. Πρώτον, για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ρόλο του στην πολιτική συνοχή. Δεν ακούσαμε πολλά πράγματα γι' αυτό. Η, το ΕΛΚ, ε, το Λαϊκό Κόμμα ε, στο Ισπανικό Κοινοβούλιο έχουμε, έχει πολλή εμπειρία για αυτό το θέμα ε, και να σας πω ότι τα κοινωνικά προβλήματα είναι τα σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι τα τεχνικά, τα τεχνικά προβλήματα και η τεχνολογία δεν είναι η προτεραιότητά μας. Τα κοινωνικά προβλήματα είναι η προτεραιότητα και λύνονται με περισσότερη Ευρώπη. Στην Ισπανία αυτό έχουμε αντιληφθεί εμείς, το Λαϊκό Κόμμα. Και μια άλλη σκέψη είναι η εξής. Οι δείκτες, μάλλον ε, οι δείκτες που χρησιμοποιούσαν πάντοτε ήταν το ΑΕΠ, ε, και κυρίως το ΑΕΠ, αλλά το ΑΕΠ εκφράζει αυτό που εκφράζει, τίποτα παραπάνω. Μέσα στο ΑΕΠ δεν υπάρχει καμία μνήμα της κοινωνίας, δεν υπάρχει καμία κοινωνική πτυχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εγκρίνει και άλλους δείκτες, όχι μόνο το ΑΕΠ. Γιατί πίσω από το ΑΕΠ κρύβονται πολλά κοινωνικά προβλήματα τα οποία το ΑΕΠ δεν μετράει. Αυτές είναι οι σκέψεις του Λαϊκού Κόμματος στην Ισπανική Βουλή. Ευχαριστώ. Ε, Ο Βίκτορ Μποστινάρου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ρουμάνο Ευρωβουλευτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι μια πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Και μην ξεχνάτε το εξή. Καταρχά, Καταλαβαίνω τις θεμητές ανησυχίες σας για την ε, μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν συστηματικά εναντίον αυτής της αιρεσιμότητας. Αλλά ούτε μία κυβέρνηση δεν υπήρχε, ούτε καν οι δικές σας, αυτών που μιλήσατε κατά. Είπαν μία κουβέντα εναντίον είναι το θεσμικό σας καθήκον να το συζητήσετε αυτό το θέμα και να καταλάβετε γιατί οι κυβερνήσεις σας συμπεριφέρθηκαν όπως συμπεριφέρθηκαν. Δεύτερη παρατήρηση. Θέλω να συζητήσουμε το Ταμείο Συνοχής, πρικοδοτημένα με 66 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 10 θα πάνε για τη διευκόλυνση ιδιώντας στην Ευρώπη. Είναι τεράστιο ποσό, αλλά τα χρήματα μπορούν να δαπανηθούν σοφρά εάν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο υπάρχει από 1η Ιανουαρίου. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τις πόλεις, για τις περιφέρειες, για τους Ευρωπαίους πολίτες σε κάθε κράτος μέλος. Και την κεντρική θέρμαση. Είναι τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο στην κεντρική Ευρώπη, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Έχουμε επιλύσει το πρόβλημα εξοικονόμησης ενέργειας αλλάζοντας τα κτίρια, ε, εξυγχρονίζοντας τα και τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Και αυτό είναι μεγάλη καινοτομία. Και, και στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για το οποίο είναι υπεύθυνος ο Γιάνν ε, Όλμπριχτ, και στο Ταμείο Συνοχής υπάρχει αυτή η μνήμα. Επίσης λύσαμε το πρόβλημα της διανομής και μεταφοράς ενέργειας, θέρμασης και ψήξης. ενέργεια τρίτης γενιάς. Επίσης, τη δυνατότητα επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα, εσείς και εμείς μαζί θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση ολιστική για όλα τα ταμεία. Μπορούμε τώρα να συνδυάσουμε τους πόρους από το, από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ταμείο Συνοχής, αν θέλουμε να πάνε αυτά τα λεφτά για τις μεταφορές, ε, την θέρμανση και την ψήξη και την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά για να αντιμετωπίσουμε ολιστικά τα ταμεία χρειαζόμαστε οι διαχειριστικές αρχές να δημιουργηθούν για να υπάρξει αυτού του τύπου η διαχείριση. Αυτή η προσέγγιση η συμπληρωματική των ε, ταμείων συνδέεται με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ούτως ώστε να σχεδιάσουμε την αρχή προγράμματα που καλύπτουν και τις δύο διαστάσεις. Και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Σας είπα από την αρχή ότι τα 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής θα δοθούν για τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρχή ήταν το μόνο που πολέμησε για να μείνουν τα 10 δισεκατομμύρια στο, ως ποσό για τα κράτη συνοχής. Και το βάλαμε αυτό και στο Γενικό Κανονισμό και στο Ταμείο Συνοχής και στη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Δηλαδή τα ποσά αυτά να παραμείνουν στο εθνικό πλαίσιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016. Αυτό ωραίο και καλό ακουγόταν, αλλά για να μπορούμε για να μπορούμε να επενδύσουμε αυτά το 15% των ποσών του Ταμείου Συνοχής χάρη στο, στη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, θα πρέπει να ετοιμάσουμε από τώρα τα προγράμματα και για την ενέργεια και για τους συντροδρόμους και για την ευρυζωνικότητα και για το φυσικό αέριο. Εάν τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση ή δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αυτό το 15% των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής σε συνοριακά προγράμματα με τα όμορα κράτη-μέλη, από 1η Πρώτου του 2017, το 15% των δικών σας κονδυλίων συνοχής θα πάνε πίσω στις Βρυξέλλες. Σας το λέω και κρούω τον κόδωνα. έχουμε βάλει μεγάλη έμφαση στην, στο διοικητικό και θεσμικό δυναμικό. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να δημιουργήσουν το δικό τους δυναμικό, ούτω ώστε να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τέτοιου τύπου προγράμματα. Αυτή ήταν η δική μας συνεισφορά. Εμείς είπαμε αυτά που είπαμε, υιοθετήσαμε τους απαραίτητους κανονισμούς και τώρα το μπαλάκι είναι στα εθνικά κοινοβούλια για να αξιολογήσουν την ετοιμότητα των, των κυβερνήσεων των κρατών μελών για να εφαρμόσουν αυτά τα προγράμματα. Τα δικά σας κοινοβούλια. Είναι δικό σας, έχετε το, εσείς το εθνικό καθήκον και το θεσμικό καθήκον, το ώστε οι αρχές στα κράτη-μέλη σας να εφαρμόσουν σωστά και έγκαιρα αυτά τα πράγματα. Τα μα μου καλά είναι, αλλά δεν πρόκειται να τα ακούσει κανένα και δεν θα δώσουν και αποτελέσματα. Έχετε μια τεράστια ευθύνη. Το Συμβούλιο μαζί με τις κυβερνήσεις σας ήταν επικεντρωμένα με μονομανία στη διακυβερνητική διάσταση και προσπαθούσαν να επιλύσουν τα προβλήματα έτσι, κυβέρνηση με κυβέρνηση, μεταξύ των κυβερνήσεων. Ενώ εμείς μαζί με την Κομισιόν καταφέραμε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι να αφήσουμε το αποτύπωμά μας. Ε, περνώντας αυτή την κοινοτική μέθοδο. Τώρα όμως που την περάσαμε αυτή την κοινοτική μέθοδο, ας την εφαρμόσουμε. Και είμαι πεπισμένος ότι οι περιφέρειές μας και οι κοινότητές μας χρειάζονται σε μια εποχή ε, σπάνιδας πόρων μια σωστή πολιτική συνοχής. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από πρώτης πρώτου του 2014 είναι έτοιμα τα κράτη-μέλη, αν όχι στην αρχή, στο τέλος του 2014. Αλλιώς θα αρχίσουν όλα να παραπονιούνται και η χώρα που θα αρχίσει τα ίδια. Είναι περίπλοκα, θέλουμε και άλλο χρόνο. Αλλά ο λαός μας, οι λαοί μας δεν έχουν υπομονή για να περιμένουν ακόμα περισσότερο. Από την Κροατία, ο Πέτερ Μπερενόβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε την ευκαιρία, έχω την ευκαιρία να μιλήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας μιλήσω για τη δική μου εμπειρία από τη δική μου χώρα, που είναι το πιο καινούριο, το πιο νέο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σας πω λίγα πράγματα για, κάποια ε, για θέματα που ακούσαμε ξανά και ξανά στη συζήτηση. Κάποιοι ομιλητές είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να επιμείνει στην δημοσιονομική πειθαρχία σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Αυτό είναι καλό κατά την απόψή μας, γιατί στην Κροατία είχαμε περιπτώσεις όπου έγιναν επενδύσεις χωρίς σαφή στρατηγική και χωρίς στόχο έγιναν εισμάτιν αυτέ οι επενδύσεις. Ακόμα και οι πιο ανεπτυγμένε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν πια την πολυτέλεια να κάνουν τέτοιου τύπου αστόχαστες επενδύσεις. Δεύτερον, κάποιο που για μας είναι αναπτυξιακή προτεραιότητα στην ε, Κροατία είναι η ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση, αυτό το πρόβλημα. Δεν έχει αρκετή ενέργεια, πρέπει να αυξήσουμε την, ενεργειακή, την ενεργειακή αποδοτικότητα, πρέπει να φτιάξουμε ενεργειακές υποδομές και οι εθνικές μας στρατηγικές συνάδουν απόλυτα με την ε, ευρωπαϊκή στρατηγική σε αυτό το τομέα. Και ελπίζουμε να υπάρξει υποστήριξη ούτως ώστε να εφαρμόσουμε αυτή τη στρατηγική. Υπάρχει επίσης το θέμα, ακούστηκε το θέμα του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στην ε, εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής συνοχής το ότι έχουν περισσότερε αρμοδιότητε για να κάνουν περισσότερα. Με βάση την εμπειρία μου και φαντάζομαι και τη δική σα, μπορούμε να συμφωνήσουμε νομίζω ότι όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι εθνικέ κυβερνήσει έχουν ένα σαφέ πλαίσιο μπροστά του, μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν. Και αυτό είναι το κοινοτικό κεκτημένο. Θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκδώσει ένα συγκεκριμένο έγγραφο που θα επιβάλλει σε όλες τις κυβερνήσεις μια νομική υποχρέωση να εμπλέκουν τα εθνικά τους κοινοβούλια στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε πραγματικά έχω δισταγμούς για το κατά πόσο μπορούμε να πείσουμε τις κυβερνήσεις μας να κάνουν κάτι τέτοιο. Χρειάζονται έτσι μια παρότρινση. αναφέρθηκε ε, το νησί Κιόρκ στην Ανατολική Αδριατική και ο σταθμός που υπάρχει για το υγροποιημένο αέριο. Ούτως να ε, είπαμε ότι πρέπει να μεγαλώσει αυτός ο σταθμός, ούτως ώστε να λαμβάνει περισσότερες ποσότητες τέτοιου αερίου και να το μεταφέρει στην ε, ενδοχώρα. Αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό για την Κροατία, αλλά είναι τέτοιου είδου προγράμματα σημαντικά για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση ο στόχο μας είναι τελικά να αποκτήσουμε ενεργειακή ανεξαρτησία. Και με τέτοια προγράμματα μπορούμε να βοηθηθούμε. Ε, η εμπειρία που έχουμε από κάποιε συμφωνίε εταιρική σχέση δεν ήταν 100% θετική. Ας το πούμε ξεκάθαρα, α είμαστε ειλικρινεί. Εμείς επειδή μπορούμε, δεν μπορούσαμε να δεχτούμε να συμφωνήσουμε με τις όμορες χώρες μας, δεν μπορούσαμε να πούμε ποια είναι η, οικονομική μας ζώνη. λαός μας, ε, γιατί δεν συμφωνούσαμε με την Ιταλία και με άλλες γειτονικέ χώρες. Είναι σημαντικό να γίνει κάτι για αυτό το πράγμα. Η Κομισιόν θα μπορούσε να πάρει μια πρωτοβουλία εκεί και να κινηθεί εξ ονόματος των ε, χωρών που θέλουν να αντλήσουν ε, χρήματα από τα ταμεία. Κάτι τέτοιο θα ήταν εποφελές ε, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Ζέλερ, Ευρωβουλευτής, ήταν εισηγητής για την τροποποίηση του κανονισμού για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Ενταφικής Συνεργασίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που αναφέρατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την περιφερειακή συνεργασία που είναι ένα νομικό μέσον για, με, την τωρινή του μορφή ε, για την επιτεύξη στόχων της πολιτικής συνοχής. Ε, και ευχαριστώ όσους συνεργάστηκαν για να γίνει. Θέλω όμως να αναφερθώ σε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί είναι καλή ε, ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν πρέπει όμως να γίνεται σποραδικά μια φορά το χρόνο, αλλά πιο συχνά και σε μεγαλύτερη σύνθεση. Γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας μας αναθέτει κοινή ευθύνη για την ευρωπαϊκή πολιτική και τα μέσα που αυτή διαθέτει. Όμως τώρα Ακόμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπραγματεύεται με το Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις δηλαδή, και από τα λόγια σας ακούω ότι η ομολογή σας είναι η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις. Οι κεντρικές ε, διοικήσεις δηλαδή εξακολουθούν να κυριαρχούν. Όμως δεν μπορεί στο Δινεκές να συνεχίσει αυτή η κατάσταση ιδιαίτερα ε, αν θέλουμε να ε, απαλείψουμε τα δημοκρατικά ελλείμματα. Εμείς είμαστε οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι και μπορούμε τα δημοκρατικά αυτά ελλείμματα να τα εξαλείψουμε. Από πολλές παρεμβάσεις σας προέκυψε επίσης ότι η κρίση στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και των περιφερειακών φορέων δεν έχει ξεπεραστεί, που δεν και χρειάζονται κοινέ προσπάθειες ούτως ώστε να βάλουμε πάλι σε, στο μονοπάτι της ευημερία τους πολίτες μας και να τους εξασφαλίσουμε καλό επίπεδο ζωής. Το θέμα είναι αν οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε μέχρι τώρα εξυπηρετούν την επίτευξη του στόχου με τα διαρθρωτικά ταμεία, την πολιτική συνοχής έχουμε δυνατότητα να βοηθήσουμε τις πιο αδύναμες περιφέρειες. Τώρα πλησιάζουμε στο τέλος του 2013 και στο τέλος της περίοδου της αναπτυξιακής 2007-2013. Ήδη τον Ιανουάριο, δηλαδή σε 6 εβδομάδες περίπου, θα πρέπει τα νέα μέσα να είναι στη διάθεσή μας για την ανάπτυξη. Στην τελευταία στιγμή καταφέραμε, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, να βρούμε μια συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και κυβερνήσεων. Οι προτάσεις της Κομισιόν αναμένονταν ήδη από το, την άνοιξη του 2011, δηλαδή επί Πολωνικής Προεδρίας. Ε, τις ελάβαμε σε 7 Οκτωβρίου του 2011 και σε ό,τι αφορά το Πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τις βασικούς κανονισμούς και τις άλλες νομοθετικές προτάσεις. Το Κοινοβούλιο αντέδρασε σχετικά γρήγορα. Τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2011 ε, είχαμε τις αποφάσεις και για το πολιετές δημοσιονομικό και για τα διαρθρωτικά ταμεία. Μετά πέρασε 1,5 χρόνος όπου διαπραγματευόμαστε και συζητούσαμε με το Συμβούλιο και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή εξευρέθη συμφωνία. Υπήρξαν συζητήσεις, ε, επισυζητήσεων, σχολαστικές συζητήσεις και πολλές φορές ε, είχαμε αντιπαραθέσεις και στους κόλπους του Συμβουλίου που δεν συμφωνούσε σχετικά με τη διαμόρφωση του κειμένου. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι ε, οι μηχανισμοί αυτοί, τα μέσα αυτά χρειάζονται για την υπέρβαση της κρίσης. Προέκυψε επίσης από τις ομιλίες ε, ότι η Κομισιόν άρχισε πλέον να διαπραγματεύεται για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, να καταρτίζει επιχειρησιακά προγράμματα, να ε, τα ελέγχει και όπως είπε πρόσωπος της Κομισιόν τώρα εξετάζουν πάλι τις εξάντε κοντισονάλιτες αυτές τις ε, εκ των προτέρων ερεσιμότητες. Ε, η θεματολογία πρέπει να επικεντρώνεται σε αυτό που αποτελεί την ευρωπαϊκή στρατηγική. Ε, ο κ. Σόμπερ ως εκπρόσωπος ε, Περιφερειακής Ένωσης λέει ότι είναι καλή η θεματική συγκέντρωση, ο κ. Ρόμπρα, αλλά χρειαζόμαστε και μια ουσιαστική ευελιξία αφού οι περιφέρειες είναι τόσο διαφορετικές μεταξύ τους. Άρα λοιπόν ενώ πρέπει να αρχίσει η δουλειά, αρχίζει άλλη συζήτηση σε σχέση με τον κανονισμό τον εφαρμοστικό. Και το ερώτημα είναι αν διαθέτουμε αυτό το χρόνο και αν από τα αποτελέσματα μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Πολλές φορές οι συνάδελφοι και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπαν ότι θα πρέπει να πιέσετε τις κυβερνήσεις ούτως ώστε να λειτουργήσουν πιο θετικά στο Συμβούλιο για να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση. Έτσι θα επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, γιατί συχνά συμβαίνει ε, το εξής μεταξύ των απαιτήσεων που υπάρχουν, μεταξύ των υφισταμένων δυνατοτήτων αλλά και της πραγματικότητας ε, το κενό να βαθαίνει όλο και περισσότερο. Έχουμε το θέμα της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. Βέβαια πρέπει να ρυθμίσουμε τη χρηματοπιστωτική αγορά. Θα πρέπει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να σταθεροποιηθούν. Δίνει πολλά λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Χρησιμοποιούνται όμως ως επιτοπλίστων για να σταθεροποιηθούν οι τράπεζες και το χρήμα το οποίο παίρνουν τόσο φθηνά δεν ε, χρησιμοποιείται για επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει εγγύησεις, χορηγεί εγγύησεις και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, χρηματοδοτικά μέσα για να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα προγράμματα και να τα αφήσει να υλοποιηθούν. Αυτά τα μέσα ως επιτοπλίστων όμως δεν αξιοποιούνται, δεν χρησιμοποιούνται και έτσι γυρίζουμε σε κύκλους και βάζουμε τρικλοποδία στον εαυτό μας. Δεν αξιοποιούμε τις υφιστάμενες δυνατότητες. Βέβαια αυτές οι εσωτερικές αδυναμίες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολουθούνται έξωθεν και πολλές φορές ε, χρησιμοποιούνται και προσφέρονται και ξένα κονδύλια. Οι Κινέζοι δίνουν τα λεφτά τους, ε, ούτως, γιατί έχουν συσσωρεύσει, συσσωρεύσει τεράστια εμπορικά ισοζύγια για να ε, κάνουν επενδύσεις. Ε, έγινε μια συνδιάσκεψη στο Βουκουρέστι με πολλά, συμμετοχή πολλών κρατών όπου οι Κινέζοι ε, προσφέρουν δισεκατομμύρια σε επιστώσεις προκειμένου να εφαρμοστεί όμως η δική τους η τεχνολογία. Ε, έχουμε τα ευρυζωνικά, τη διαλειτουργικότητα, τα ενιαία τεχνικά πρότυπα. Η Κίνα ε, λέει ότι αν αγοράσετε τα τρένα υψηλής ταχύτητας ε, θα κάνουμε επενδύσεις. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι τα προβλήματα δεν γίνονται λιγότερα. Αλλά Λύση μπορούμε να βρούμε μόνο αν ενισχύσουμε τη δικτύωση μεταξύ μας, τα δίκτυα και πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα. Ο κύριος Έκης από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πολλές φορές ε, κανείς ετοιμάζεται να ετοιμάζει μια ομιλία για τέτοιου είδους συναντήσεις και ξαφνικά του έρχονται καινούριε ε, ιδέες. Η Ουγγαρία υπέβαλε το έγγραφό της για την ε, εταιρική σχέση και έλαβε θετικά σχόλια. Και κατόπιν έγινε πολλή συζήτηση και στη χώρα μας. Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την ε, Ουγγρική Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης το Μάρτιο 2013 και ταυτόχρονα ε, τον ε, θεσμό του διαμεσολαβητή για το μέλλον. Νομίζω ότι χρειάζεται ένας διαμεσολαβητής στην νομοθεσία προκειμένου να ελέγχει και ενδεχομένω να βάζει και βέτο όταν δεν ε, λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα της επόμενης ή των επόμενων γενιών. Στην Αυστρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία ε, και σε άλλες χώρες ε, δημιουργούνται ταυτόχρονα δίκτυα ενέργειας και, όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με τους κατάλληλους κανόνες. Στη Γερμανία υπάρχει ένα θέμα κανόνων. Το Ουγγρικό Κοινοβούλιο από την άλλη μεριά για αυτό το λόγο ε, υιοθέτησε τη δική του στρατηγική και τους δικούς του κανόνες. Ε, επίσης έχουμε και στρατηγική περιβαλλοντικής, ε, ναι, περιβάλλοντος, ανάπτυξης της υπαίθρου κλπ. Πάντοτε κοιτώντας το μέλλον, κοιτώντας το αύριο για να εξασφαλίσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ουγγαρίας θα είναι πιο ισχυρές και ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Το 2014 ξεκινάει μια καινούργια εποχή με αποκεντρωμένα όργανα λήψης αποφάσεων. Γιατί δεν υπάρχουν δύο περιφέρειες ίδιες μεταξύ τους στον κόσμο. Πρέπει λοιπόν οι πόλεις, οι νομοί, τα διοικητικά διαμερίσματα, οι περιφέρειες να ε, πούν ποιες είναι οι ανάγκες τους. Στη Βουδαπέστη έγινε πριν από κάποιο καιρό μια συνάντηση όπου ε, Ρουμανοί, Σέρβοι και Γερμανοί βουλευτές μας επισκέφθηκαν ε, κατόπιν ε, πρωτοβουλίας Γερμανικού Ινστιτούτου και εκεί μιλούσαμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή. σε ε, πάρτε τα γενετικά τροποποιημένα ε, ε του γενετικά τροποποιημένου σπόρους. Ε, ναι. Αν δεν αναπτυχθεί σωστά η κάμπια θα βγει ποτέ πεταλούδα, έτσι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς. <clears throat> αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε. Ε, θα πρέπει να δούμε ε, να προσπίσουμε την, από, ανταγωνιστικότητά μας έναντι της Κίνας των ΗΠΑ και άλλων. Ο κ. Μπαρόσο είπε ότι η οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης κινδυνεύει σήμερα εξαιτίας ε, του, του, του υψηλού κόστου των δημοσίων υπηρεσιών. Πρέπει να δούμε λοιπόν το ξανά το θέμα της ενέργειας, της διασύνδεσης των δικτύων, του κανονιστικού πλαισίου και της εταιρικής σχέσης. Σε θέματα ανταγωνιστικότητας, ε, θα έπρεπε να έχουμε όλοι μια κοινή φωνή. Οι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε μια αποτελεσματική συνεργασία και μια βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα. Ιδιαίτερα τώρα περνάω μια εποχή κρίση. Ευχαριστώ. From the European Parliament, the last speakers from Spain. Η Μαρία Ριγόιν Πέρες, τελευταία ομιλήτρια πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, θα ήθελα οι διερμηνείς να μείνουν μαζί μας γιατί θέλουμε να ακούσουμε και τους, ε, τους ομιλητές του πάνελ. Ε, κύριε Ριγκόγεν, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη και να απαντήσω και σε ορισμένα από τα σχόλια τα οποία έγιναν. Α, νομίζω ότι τελικά μας απασχολούν τα ίδια θέματα όλους, αλλά ο καθένας έχει τις ευθύνες του στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Εμείς στο ευρωπαϊκό επίπεδο και οι εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων στο εθνικό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να απαντούν και να ανταποκρίνονται τις αρμοδιότητες τους σε εθνικό επίπεδο και εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς τέτοιου είδους ε, συνεδρία συναντήσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες διότι συντονιζόμαστε και ακούει ο ένας τη φωνή του άλλου. Τα παράπονα στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, που ε, τα παράπονα που εξέφερε για παράδειγμα ο Ισπανός εκπρόσωπος από τη Γερουσία να τον ενημερώσω ότι η συνοχή είναι επένδυση σε ανθρώπους για να αναπτυχθούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή, ε, ανάπτυξης, ε, η αυτή η Επιτροπή ε, ζήτησε το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να πάρει το 25%. Στις συζητήσεις που έγιναν <clears throat> για τον οριζόντιο κανονισμό το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 23,1% από το Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο ε, η Ισπανία εκπροσωπήθηκε από την κυβέρνησή της. Συνεπώς, ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του εκεί που πρέπει. Τώρα, στον ε, Γενικό Διευθυντή να πω το εξής για την εφαρμογή των ταμείων. Τα, τους, ε, τους τελευταίους μήνες εγώ συμμετείχα σε πολλές συναντήσεις στην Ισπανία και όλοι μου επαναλαμβάνουν το ίδιο. Δεν υπάρχει έλλειμμα, υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης. Δεν ξέρω αν ε, η Γενική Διάθεση Regio έχει σκοπό να αυξήσει το προσωπικό ε, που διαχειρίζεται τα ταμεία, αλλά αυτή τη στιγμή υφίσταται έλλειψη ενημέρωσης για, την, ε, για τις κυβερνήσεις. Ξέρω ότι εξαιτία τη αλλαγή νομοθεσία έχουν πληγεί τη δουλειά. Όμω με ρωτάνε τι θα γίνει με το άρθρο 5. Τι πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δηλαδή είναι πολύ εύκολο να τους ενημερώσουμε για τα χρονοδιαγράμματα. Από πότε θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι, αρχές, οι συμφωνίες ε, και πότε θα πρέπει να είναι έτοιμα τα επιχειρησιακά σχέδια. Και ένα τελευταίο σχόλιο για την Δανέζα συνάλφο γιατί μου το προκάλεσε πραγματικά. Πολύ καλές οι προθέσεις της, Καταλαβαίνω, όλοι θα θέλαμε να έχουμε μια τέτοιου είδου σχέση με, όλοι μέσα σε μια κοινότητα να έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους, όλοι να υποφελούνται από τα μέτρα και οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται, αλλά δυστυχώς η παγκοσμιοποίηση μας αφορά όλους και ε, είναι ε, απόλυτα ε, αναπόφευκτες οι φούσκες. Ε, οι οποίες σκάνε κιόλα. Η χρηματοπιστωτική κρίση έγινε μακροοικονομική κρίση και επεκτάθηκε σε όλο τον πλανήτη. Ήταν το αποτέλεσμα ενός ντόμινο που επηρέασε όλους. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν να απαντήσει πρώτη. Και οποιοδήποτε από τους ομιλητές του πάνελ θέλει να απαντήσει, πολύ ευχαρίστως. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις για τα σχόλιά σας. Ακούστηκαν τόσα πολλά σχόλια, τόσες παρεμβάσεις που είναι δύσκολο να απαντήσω σε όλα. Θα προσπαθήσω να είμαι συγκεκριμένος, ανοιχτό, ανοιχτός, αλλά και λίγο σκληρός. Να σας πω πού βρισκόμαστε. Τα επενδυτικά και διαφορετικά ταμεία για την επόμενη περίοδο είναι πολύ σημαντική ε, πηγή δημοσίων επενδύσεων για τις περισσότερες χώρες. Ε, και για ορισμένε περιφέρειε είναι και η μοναδική πηγή. Όταν κάνει επενδύσει, θα πρέπει καταρχά να κάνει μια ανάλυση των αναγκών, θα πρέπει να δει τι αποτελέσματα θε να πετύχει με αυτέ τι επενδύσει και μόνο τότε να πει ποια θα είναι τα συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία θα επενδύσει. Και δηλαδή ποια προγράμματα τελικά θα υποστηρίξει για να υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα. Αυτό είναι κάτι που έλειπε, γι' αυτό έχουμε νέου κανονισμού, οι οποίοι είναι πολύ πιο υγιεί και σωστή και λαμβάνουν υπόψη ε, αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για αυτά, για αυτού τους κανονισμού. Είναι η μισή δουλειά μα αυτή. Έγινε δουλειά από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Τώρα έχουμε του κανονισμού και μια και του έχουμε υπάρχει μια τεράστια ευθύνη σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Γιατί πρόκειται για επιμερισμένη διαχείριση. Και βλέπω που μπαίνει και η ευθύνη των κρατών μελών. Είχαμε τις τις ίδιες ευκαιρίες για όλα τα κράτη-μέλη. Όταν πριν από 1,5 χρόνο ε, καλέσαμε τα κράτη-μέλη να έρθουν, η πρόεδρος διακόπτη, γιατί λέει ότι οι διερμηνείς πρέπει να φύγουν ως ονούπο. Υπάρχει ένας ε, κώδικας διοντολογίας. Ε, όσοι θα συνεχίσουν ε, θα πρέπει να μας ακούσουν αγγλικά. Θα συνεχίσουμε αγγλικά δηλαδή, χωρίς τους διερμηνείς. Εγώ θέλω να πω συνεχίζει ο κύριος Πόπενς, ότι δουλέψαμε πολύ. Και ο νέος κανονισμός θα βάλει μεγάλο άχθος ε, στο εθνικό επίπεδο για να σχεδιάσουν ε, τα σωστά εργαλεία, έγγραφα κτλ. Όχι για να μας ευχαριστήσετε, αλλά γιατί αν θέλετε να κάνετε σωστές επενδύσεις πρέπει να τα έχετε όλα αυτά. Μόνο 14 κράτη-μέλη σήμερα μας έδωσαν σχόλια πλήρη και ελπίζω τα υπόλοιπα κάτι μελη που δεν έχουν κάνει κάτι τέτοιο ε, θα έχουν όριμες συμφωνίες εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράμματα. Ε, ή μάλλον αυτά τα 14 που έχουν υποβάλει τα, τα σχόλιά τους. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα υπόλοιπα 14. Δεν θέλω να ονοματίσω και να στυλιτεύσω κανένα εδώ, αλλά είναι λογικό τα εθνικά κοινοβούλια να επιστρέψουν στις κυβερνήσεις και να τους πούν «Μα πού βρίσκεστε σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις, υπάρχουν οι επενδύσεις, ε, τελειώνει ο διάλογος και θα ετοιμαστούν οι εκθέσεις». Δηλαδή θα μπούμε στην ε, επίσημη τελική φάση και εκεί σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε, επίσης θα πρέπει να γίνει α, και όλη η δουλειά από την αρχή με τα υπόλοιπα 14 κρατημέλη που δεν έχουν ακόμα δώσει σημεία ζωής όταν Ξέρετε ότι κλείνει όμως, όπως σας είπα, ο άτυπος διάλογος. Το θέμα της συγκέντρωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η συνταγή με το ΚΕΚ καλή είναι. Το θέμα δεν είναι τι μυρωδικά θα βάλεις. Το θέμα είναι να έχουμε μια καλή βάση για το ΚΕΙ και ε, να έχεις περισσότερο αλεύρι για την ουσία, όχι περισσότερα έτσι, μπαχαρικά. Πρέπει να βρούμε τρόπους για να υποστηρίξουμε, υποστηρίξουμε μέσω των ταμείων τις επενδύσεις αυτές, ούτως ώστε να το φτιάξουμε αυτό το κέικ τέλος πάντων. Ε, έχουμε τις, εκ των προτέρων, ε, την πρωτόν ερεσιμότητα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε από τα ταμεία στην ε, οικοδόμηση διοικητικού δυναμικού, αλλά πρέπει να δούμε μαζί με τα κράτη-μέλη σε ποιους τομείς. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά ακόμα. Εγώ πήγα στην ε, Ισπανία για να εξηγήσω τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη νέα περίοδο. Έγραψα στα κράτη-μέλη πριν από 1,5 χρόνο, όταν υποβλήθηκαν ε, έγγραφα στα κράτη-μέλη. Τώρα είναι η στιγμή να κινητοποιηθούμε σε όλα τα επίπεδα, γιατί πρόκειται για μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Είναι η νέα προσέγγιση Πρέπει να υπάρχει εθνικός διάλογος ε, με τη συμμετοχή του περιφερειακού επίπεδου και του τοπικού επίπεδου. Λυπούμαστε, αλλά πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Οι διερμηνείς σταματούν εδώ και σας καληνυχτήσουν. Γεια σας. Together with that. So it's very important to mobilize now forces at national level. The window is still open for informal dialogue